που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 28 Νοεμβρίου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη είχε τη δυνατότητα να συζητήσει το θέμα αυτό με την Οικονομική Επιτροπή στις 2 Δεκεμβρίου. Προσβλέπω σε περαιτέρω συζήτηση του σημαντικού θέματος μαζί σας σήμερα και στο μέλλον. Θα ξεκινήσω επενθυμίζοντας ότι η οικονομική και η χρηματοστατική κρίση έδειξε ότι είχαμε μεγάλες αδυναμίες στην αρχική οικονομική και νομισματική ένωση και το σύστημα η Ευρωπαϊκή Ένωση αντέδρασε σε διάφορα μέτωπα. Η δράση πραγματικά ήταν εντυπωσιακή, κυρίως όταν συγκριθεί με αυτό που εθεωρεί το εφικτό πριν από κάποια χρόνια. Η Ευρωζώνη ενισχύθηκε σημαντικά με μόνιμο τείχος προστασίας στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας εξασφαλίζεται έτσι η οικονομική σταθερότητα. Δημιουργήσαμε μια τραπεζική ένωση για να αντιμετωπίσουμε τον κατακαιρματισμό του οικονομικού τομέα και να διευκολύνουμε την πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Εν τέλει ενισχύσαμε την οικονομική μας διακυβέρνηση ώστε να ενισχύσουμε την οικονομικό και δημοσιονομικό συντονισμό. Ε, το εξάπτυχο πακέτο και το δίκτυχο ε, πακέτο θα ενισχύσουν την οικονομική διακυβέρνηση, θα ενισχύσουν την εποπτεία του προπολογισμού στα πλαίσια του Συμφώνου Σταθερότητα και Ανάπτυξη. Ο έλεγχο αφορά και την μακροοικονομική ανισορροπία και αντιμετωπίζει και τα προβλήματα ανισορροπίων σε διάφορες χώρες και έχουμε και κωδικοποίηση νομοθεσίας ολοκληρωμένου οικονομικού ε, και χρηματοστικού ελέγχου στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμείνου. Σύμφωνα με τι νομικέ απαιτήσει στα διάφορα νομοθετήματα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ολοκλήρωσε την αναθεώρηση των νέων μέσων που θεσπίστηκαν. Εν γέννη, η αναθεώρηση επιβάλλει να αξιολογήσουμε τρία στοιχεία του εξάπτυχου πακέτου και του δίπτυχου. Ε, θέλουμε να βρούμε τους διάφορου σε ποιο βαθμό οι νέοι κανόνες ήταν αποτελεσματικοί για την επίτευξη των στόχων. Δεύτερον, πρέπει να αποφύγουμε τον αντίκτυπο των κανόνων. Πρέπει να έχουμε καλύτερο συντονισμό για τις οικονομικές πολιτικές και να ενισχυθούν τους κανόνες και θέλουμε οι κανόνες αυτές να βελτιώσουν και να στηρίξουν την οικονομική εποπτεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε πολύ περιορισμένο χρονικό διάστημα από όταν είχε τεθεί σε ισχύ. Η εμπειρία όσον αφορά το νέο σύστημα είναι περιορισμένη και διάφορα συγκεκριμένα εργαλεία δεν έχουν δοκιμαστεί ακόμα. Αφορά πιο συγκεκριμένα το σύστημα, τη ε, διαδικασία των υπερβολικών ισορροπιών και το σύστημα μέχρι τώρα εφαρμόστηκε σε συγκεκριμένε οικονομικέ συνθήκε κατά τη διάρκεια και μετά την σοβαρή κρίση αυτό περιόρισε τις δυνατότητε να δούμε αν είναι αποτελεσματικό το σύστημα όσον αφορά την πρόληψη. Για αυτούς τους λόγους η αναθεώρηση που ε, δημοσίευσε τον Νοέμβριο η ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι σύντομη ε, και αποτιμά την χρήση του συστήματος, δηλαδή από το φθινόπωρο 2011 για το εξάπτυχο και από το 2014 για το δίπτυχο σύστημα. Λοιπόν, για τις μακρονόμιες ισορροπίες και για το πλαίσιο λοιπόν των χωρών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά χρηματοδοτική ισορροπία έχουμε σαν στόχο. Αναφέρονται και διασυνδέσεις μεταξύ των διαφόρων στοιχείων. Η αναθεώρηση, η έκθεση αναφέρει κάποιες ε, βελτιώσεις που έχουν επιφέρει ε, μεταρρυθμίσεις στο δίπτυχο και ε, εξάπτυχο τομέα. Βελτιώθηκε η οικονομική διακυβέρνηση και έχει επιτευχθεί πρόοδος όσον αφορά την εξυγίανση των δημοσιονομικών και την διόρθωση των μακροοικονομικών ισορροπιών. Και τέλος εντοπίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάποιους τομείς για ενδεχόμενες βελτιώσεις αφορά τον περίπλοκο χαρακτήρα του συστήματος όσον αφορά την αλληλεπικάλυψη διαφόρων συστημάτων και τον περίπλοκο χαρακτήρα κάποιων συγκεκριμένων μέσων αυτών καθεαυτών όπως στο Σύμφωνο σταθερότητα και Ανάπτυξης. Το περίπλοκος χαρακτήρας μπορούσε να δημιουργήσει προβλήματα για την εφαρμογή και τη διαφάνεια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει σε αξιολόγηση που δείχνει ότι υπάρχει ανάγκη για αύξηση των μεταρρυθμίσεων που πρέπει να γίνουν στα κράτη-μέλη και έτσι θα μπορούσαμε με τι μεταρρυθμίσεις να προχωρήσουν πιο γρήγορα και να ακολουθηθούν οι συστάσει του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για τι μεταρρυθμίσει. Έτσι, θα είχαμε βελτιωμένα αποτελεσμένα για την ανάπτυξη, για τη σύγκληση και την εξάλληψη ανισορροπιών. Και η έκθεση αναφέρει την ανάγκη περαιτέρω συμμετοχή των Εθνικών Κοινοβουλίων και των εμπλεκομένων Φορέων, ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη νομιμότητα και λογοδοσία. Το σύστημα οικονομική διακυβερνήσεω μπορεί να πετύχει το πλήρε του δυναμικό μόνο αν συμμετέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορεί και τον στερνιστούν, όπω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που είναι βασικό θεσμικό όργανο που εξασφαλίζει την δημοκρατική νομιμότητα και τη λογοδοσία ε, των οικονομικών πολιτικών και των σχετικών αποφάσεων στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι το έγγραφο αυτό είναι μια καλή αφετηρία και βάση για διάλογο και για να συζητηθούν οι ενδεδειγμένε πορείε στο μέλλον. Ε, κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, προσβλέπω στην ακούσω τι σα. Σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Τώρα θα πάρουν τον λόγο οι μιλητές εξ των πολιτικών ομάδων. Κύριος Μπάλτς, ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Ως Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα βεβαίως χαιρετίζουμε την σημερινή συζήτηση. Υποστηρίζουμε την Κομισιόν καθώς βλέπουμε την ε, τωρινή νομοθεσία για το διπλό και το εξοπλό πακέτο θετικά και βεβαίως σιγά σιγά η κατάσταση όσον αφορά τα ελλείμματα των χωρών βελτιώνεται. Βεβαίως ε, σωστό είναι το ότι ζητείται επιτέλους να γίνουν και οι μεταρρυθμίσεις οι οποίες καθυστερούν στα κράτη-μέλη και υποστηρίζουμε την Κομισιόν όταν λέει πως το Σύμφωνο Σταθερότητας ε, και Ανάπτυξης έχει και μέλλον. Αυτό σημαίνει βεβαίως πως θα πρέπει να εφαρμόσουμε πρώτα απ' όλα τους υφιστάμενους κανόνες. Ε, το σύμφωνο αυτό είναι η αφετηρία για μια ε, ανταγωνιστική ευρωπαϊκή οικονομία. Και βεβαίως ε, δεν έχει κανένα νόημα να χαλαρώσουμε τώρα το σύμφωνο. Αντιθέτως έτσι θα αρχίσουμε να κάνουμε τους αριθμούς ε, ό,τι θέλουμε και δεν είναι σωστό να λέμε πως εμποδίζει την ανάπτυξη των κρατών μελών. Δεν είναι εμπόδιο στην ανάπτυξη το Σύμφωνο Σταθερότητας, απλά υπενθυμίζει στα κράτη-μέλη τις υποχρεώσεις τους να έχουν βιώσιμους και αποτελεσματικούς προς ανατολισμένους προς το μέλλον. Οπωσδήποτε αυτές είναι αλήθειες δυσάρεστες και δεν θα δημιουργηθεί θετικό ε, κλίμα για τους επενδυτές εάν δεν γίνουν ταυτόχρονα και οι μεταρρυθμίσεις. Η αξιοπιστία, κυρίες και κύριοι του συμφώνου, δεν επιτρέπεται να υπονομεύεται. Δεν πρέπει να υπάρχουν διαφορές ε, μεταξύ μεγάλων και μικρών κρατών και αναμένουμε από την Κομισιόν να κινείται πάντα προς το συμφέρον της Ευρώπης και να πει τα πράγματα όπως έχουν στα κάτι μέλη τα οποία καθυστερούν. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και εγώ για τους σοσιαλδημοκράτες. Κυρία Μπέρες έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Αντιπρόεδρε, ιδού το πρώτο ραντεβού αυτής της θητείας για να συζητήσουμε το σημαντικό αυτό θέμα που είναι το θέμα της οικονομικής διακυβέρνησης. Κατά τη διάρκεια της ε, προηγούμενης θητείας κάναμε ένα βήμα ανεπροηγουμένου όσον αφορά τον τραπεζικό τομέα με τη δημιουργία της Τραπεζικής Ένωσης. Το ραντεβού που, στο οποίο βρισκόμαστε τώρα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι η ευκαιρία να εφαρμόσουμε αυτό που θα επιτρέψει όχι μόνο να ξεπεράσουμε τη χρηματοδοτική κρίση, αλλά καθώς να μην μπούμε σε μια κρίση της πολιτικής ένωσης. Γι' αυτό το εργοτάξιο που δημιουργήσαμε εδώ είναι πάρα πολύ σημαντικό και μεγάλο όταν παρουσιάσατε τον απολογισμό ε, του Six και του Twin Pack, σαν νομοθέτες είχαμε θέσει ένα σημείο συνάντησης. Αυτό όμως δεν μπορεί να είναι απλώς για να γίνει αυτή η παρουσίαση που κάνατε, που είναι σύντομη και αναφέρει τα πραγματικά στοιχεία και που αγνοεί την κατάσταση ε, ε, του, του του αποπληθωρισμού και την πολύ χαμηλή ανάπτυξη της Ευρωζώνης και της Ένωσης. Ε, πρέπει να αναγνωρίσω ότι την ίδια μέρα δημοσίευσατε ένα έγγραφο που θεώρησα ότι δείχνει ε, καλύτερες προπτικές με την ετήσια εξέταση ανάπτυξης που αναγνωρίζει σοβαρότητα της καταστάσεως και κυρίως σοβαρότητα της ε, κοινωνικής κρίσης η οποία τονίζει και την προσφορά και τη ζήτηση που δέχεται την ύπαρξη ελλείψεως επενδύσεων και τον κίνδυνο ε, προβλημάτων σε διάφορους τομείς και καλεί τα κράτη-μέλη που έχουν δημοσιονομικό περιθώριο λιγμών να χρησιμοποιήσουν τα περιθώρια και τα αποθέματα. Όσον αφορά την πολυμερή διάσταση του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, ε, αναφέρεστε στην ανάγκη να τεθεί σωστή προοπτική όσον αφορά τι οικονομίε των κρατών μελών. Δυστυχώ, με κάποιο τρόπο έχω την εντύπωση ότι αυτό το πνεύμα και αυτή η προσέγγιση δεν αντικατοπτρίζεται στην αξιολόγησή σα όσον αφορά το six pack και το twin pack. Είπατε ότι δοκιμάστηκαν όλα αυτά σε κανονικό χρονικό διάστημα. Είναι κανονικό, διότι αυτοί οι κανόνε υιοθετήθηκαν ενώ δεν ήμασταν σε κανονικού καιρού για να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση που ήταν ασυνήθι. Ε, το αποτέλεσμα προφανώ δεν υπάρχει. Η συζήτηση που ανοίγεται παρόλα αυτά είναι πολυδιάστατη και θα πρέπει να φροντίσουμε να μπούμε εις βάθος. Όταν αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων τον Ιούνιο έθεσαν ραντεβού για το τέλος του έτους για να γίνει αξιολόγηση των δίπτυχων και εξάπτυχων μέτρων, ανέθεσαν και μια εντολή για να καθοριστεί το περιθώριο ευελιξίας της οικονομικής διακυβέρνησης. Και εκεί σας περιμένουμε, ελπίζουμε το έγγραφο που θα θέσετε επιτάπητος, ε, δεν θα καθορίσει νέους κανόνες, αλλά θα επιτρέψει να περάσουμε από τη λογική των αυστηρών κανόνων σε πραγματική καθοδήγηση οικονομικής πολιτικής, που δεν είναι τα ίδια πράγματα. Από ό,τι καταλαβαίνω, πολλοί ε, θέλουν να υπάρχουν κανόνες. Και εμείς θέλουμε τους κανόνες. Αναγνωρίζουμε όμως τα όρια των κανόνων όταν δεν μπορούν να εφαρμόζονται, όταν εμποδίζουν την κυριαρχία των κρατών μελών και ευνοούν να δημιουργείται ένα συνέστημα αντιευρωπαϊκό όταν είναι πάρα πολύ περίπλοκοι κανόνε για να επιτρέψουν να τι εστερνιστούν. Το όνομα που αναφέρεται, την ιδιοκτησία των κρατών. Περιμένουμε λοιπόν ε, με αυτή την ερμηνεία σα τη δυνατότητα να υπάρξει ευελιξία και πάνω απ' όλα γνωρίζουμε ότι ο δικό χάρτη είναι εκ νέου ανοιχτό για την περίφημη έκθεση ε, περιπτώσεων που εκεί θέλει να παίξει πλήρω το ρόλο του το Ευρωκοινοβούλιο, διότι όλο ο κόσμο το λέει. Εάν δεν προχωρήσουμε μαζί όσον αφορά την οικονομική διακυβέρνηση, η Ευρώπη τελικά ε, της τελευταίας ευκαιρίας είναι εδώ, είναι αυτή που είναι, αλλιώ θα διαλυθεί. Και έναντι του παγώματος που βλέπουμε συζητήσει μεταξύ κρατών μελών, ε, ε, λοιπόν, πιστεύουμε ότι θα πρέπει να ξαναρχίσουμε τις προσπάθειες, να ξαναρχίσουμε να κουβεντιάζουμε κανονικά, να συνεννοούμεθα αμοιβαία και σε αυτή την κατάσταση ε, περιμένετε να ακούσετε καλές ιδέες από το Κοινοβούλιο, να δείξει καλή βούληση το Συμβούλιο και ελπίζουμε όλα αυτά τελικά να συμπέσουν. Ευχαριστώ. ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο έχει το λόγο Κυρία Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, το χαιρετίζω ότι διεξάγεται σήμερα αυτή η συζήτηση. Μια συζήτηση για τα, ε, τις εξάπτυχες και δίπτυχες ε, ρυθμίσεις. Είναι μια συζήτηση για την επιτυχία ή όχι της ε, οικονομικής διακυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αν το δει κανείς υπό αυτό το εύρος είναι προφανές ε, ότι αυτή η συζήτηση είναι μια συζήτηση για την αποτυχία τέτοιου είδους διακυβέρνησης. Στην αρχή είχαμε κανονισμούς που ήταν σαφείς, εύληπτοι, και διαφανίσα ότι δεν θα υπήρχε πάνω από 60% χρέωση και ότι δεν θα υπήρχε ε, υπερβολικό έλλειμμα και ότι σε σχέση με την αρχή αλληλεγγύης ο κάθε κράτος θα ήταν υπεύθυνο για τα χρέη του και κανένα κράτος δεν θα υπομιζόταν χρέη άλλου, άλλου κράτους. Αυτοί οι κανόνες τώρα δεν έχουν πλέον υπόσταση. Απαμβλήθηκαν μέσα στην ε, μεταρρύθμιση του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης και αντικαταστάθηκαν από πιο περίπλοκους κανόνες με λιγότερη διαφάνεια όσον αφορά διαρθρωτικό έλλειμμα που νομίζω ότι οι λιγότεροι ευρωβουλευτές μπορούν να κατανοήσουν περί τίνο πρόκειται. Αυτά τα διαρθρωτικά έλλειμματα θα έπρεπε ετήσια να μειωθούν κατά 0,5% ετήσια και για κράτη που βρίσκονται υπό ιδιαίτερη αντιμετώπιση 0,8%. Δεν είδαμε να γίνεται κάτι τέτοιο. Η ε, μείωση των διαρθρωτικών αυτών ελλειμμάτων σε πολύ μικρά βήματα υλοποιείται σε πολύ μεγάλη απόσταση από το, από το το 2010 και το σημαντικό στοιχείο του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, η αρχή της μη ανάληψης χρεών διεράγει, παραβιάστηκε και δημιουργήθηκε μια κατάσταση όπου νέα χρέη θα μπορούσαν να δημιουργηθούν που δεν θα συνυπολογιζόντουσαν στα κράτη-μέλη όσον αφορά τους, τα δύο συστήματα. Υιοθετήθηκαν οι ρυθμίσεις των εξαπλών και διπλών ρυθμίσεων. Έχουμε ένα πολύ περίπλοκο τώρα σύστημα scoreboards καταλόγων, πινάκων επιδόσεων και όλα αυτά είναι πολύ δύσκολο να γίνουν κατανοητά. Υπάρχει λοιπόν αυθαιρεσία, κυρίε και κύριοι. Είναι η λανθασμένη πορεία αυτή που ακολουθούμε. Όλα γίνονται πιο αδιαφανή, πιο περίπλοκα, πιο ασίδατα και ανοίγουν δυνατότητες για κράτη να συνεχίσουν να δρούν ανυπεύθυνα όσον αφορά την διακυβέρνηση των οικονομικών τους, όπως στη Γαλλία πρόσφατα. Πρέπει να επανέλθουμε στην απλή ρύθμιση, δηλαδή τη μη ε, ε ανάληψη χρεών όσον αφορά την αλληλεγγύη. Κάθε κράτος ε, θα έχει τα δικά του κυριαρχικά δικαιώματα και θα πρέπει έτσι να τα ε, εκτελεί και να τα υλοποιεί ώστε να είναι υπεύθυνο. Το κράτος αυτό και μόνο αυτό το κράτος ε, θα πληρώνει τα χρέη του και όχι άλλοι. Δεν, δεν χρειαζόμαστε κάτι ξεχωριστό γι' αυτό, ούτε κάποιε συστάσει. Μπορούμε να επικεντρωθούμε σε αυτό, να υπενθυμίσουμε σε αυτά τα κράτη ότι τα χρέη αυτών των, κρεών, αυτών των κρατών μόνο από αυτά τα κράτη θα αναλαμβάνονται και όχι από άλλου για να ξεπληρωθούν. Αυτό θα υπαρκεί πλήρω ε, ω κίνητρο, ώστε στην ζώνη ευρώ να μπορέσουμε να επανέλθουμε στην πορεία τη συνετή, τη συνετού διακυβέρνηση. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ της τώρα, Φαν Χόιζεν παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Σήμερα συζητάμε την αξιολόγηση του λεγόμενου διπλού και εξαπλού πακέτου. Πακέτα μέτρων τα οποία εγκρίθηκαν τα προηγούμενα χρόνια για να διευρυνθεί το σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης. Η αξιολόγηση της Κομισιόν κάνει μια ωραία ανάλυση αλλά αποφεύγει τα σημαντικότερα σημεία συζήτησης. Δηλαδή το εάν και κατά πόσον θα πρέπει να επιδεικνύεται κάποια ευελιξία στους κανόνες του προϋπολογισμού. Η Κομισιόν λέει εδώ πέρα πως θα τοποθετηθεί τον Ιανουάριο. Οπότε μπορώ να βασιστώ μόνο σε αυτά τα οποία είδαμε ως σημάδια τις προηγούμενες ε, εβδομάδες, τα οποία δεν είναι ιδιαίτερα θετικά. Ο ίδιος ο πρόεδρος Γιούνκερ δήλωσε σε μια γαλλική εφημερίδα πως η Κομισιόν θεωρεί τους κανόνες του προπολογισμού και την εφαρμογή τους ως μια πολιτική απόφαση. Μπορεί ο καθένας νομίζω να εκτιμήσει το που ε, θα οδηγήσει αυτό. Εν τω μεταξύ αυτά τα οποία συζητάμε καθορίστηκαν πριν από ένα μόλις έτος το εξαπλώκιστο διπλό πακέτο και στην δικιά της αξιολόγηση η Κομισιόν λέει πως ε, επιτρέπεται να υπάρξει μια ελαστικότητα μόνο όταν μια χώρα έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά με τις μεταρρυθμίσεις. Όσον αφορά την αξιολόγηση του γαλλικού προϋπολογισμού για το 2015, τον προηγούμενο μήνα, ξεκαθάρισε η Κομισιόν πως η Γαλλία δεν έχει κάνει αρκετά για να συμμαζέψει τον προϋπολογισμό και την οικονομία της. Και μάλιστα μας ε, λέει η Κομισιόν πως ε, αυτό δεν βασίζεται σε αυτά τα οποία είχαμε συναποφασίσει. Τα πρώτα δεκα χρόνια λοιπόν του ευρώ έδειξαν το τι γίνεται εάν γίνονται οι κανόνε του Συμφώνου σταθερότητα αντικείμενο πολιτικού παιχνιδιού. Αυτό το οποίο χρειαζόμαστε λοιπόν τώρα δεν είναι περισσότερη πολιτική και περισσότερη ευελιξία και περισσότερη διακριτική ευκαιρία. Ανταυτού θα πρέπει το νέο ε, αυτό επενδυτικό σχέδιο να χρησιμοποιηθεί για να ενισχυθούν ακριβώς οι κανόνες και η εφαρμογή τους οι χώρες οι οποίες έχουν εφαρμόσει τις περισσότερες από τις συγκεκριμένες συστάσεις χώρα να λάβουν περισσότερη χρηματοδότηση έτσι ώστε να μην υπάρχει μόνο αν θέλετε μια ποινή αλλά και μια ανταμοιβή αυτών οι οποίοι τα πάνε καλά. Κάτι τέτοιο είναι τίμιο, ξεκάθαρο και αποτελεσματικό και έτσι θα ενισχύσουμε την εμπιστοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και για το ότι μείνατε εντό του χρόνου. Κύριε Ματίας έχει το χρόνο. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Επίτροπε, οποιαδήποτε αξιολόγηση για την οικονομική διακυβέρνηση θα έπρεπε να ξεκινάει από ένα πράγμα πολύ απλό και σοβαρό. Ότι απέτυχε δηλαδή. Απέτυχε. Οι νέοι κανονισμοί δεν ήταν αποτελεσματικοί. Διότι για την οικονομική πολιτική είχαμε περισσότερη ανεργία, λιγότερη ανάπτυξη, περισσότερε ανισορροπίε και δεν υπήρξε καμία συνεπής ε, διακυβέρνηση. Η οικονομική πρόταση λοιπόν ήταν αποτυχημένη. Είναι για τα σκουπίδια, για τον κάλαθο των αχρήστων και για το να ξαναξεκινήσει εκ νέου θα έπρεπε να ξαναξεκινήσουμε από μηδενικού σημείου για να διορθώσουμε τα πράγματα. Πρέπει να γνωρίζουμε ποιες, είναι οι τελικοί στόχοι με χειροπιασ... χειροπιαστά αποτελέσματα. Ελέγχθηκε το χρέος. Όχι. Αυξήθηκε. Ελέγχθηκε το έλλειμμα. Όχι. Απολύ... Αποτύχαμε και σε αυτό το επίπεδο. Σε σχέση με την ανάκαμψη αποτύχαμε. Υπάρχουν περισσότερες ανισοκομίε. Να μειωθούν οι δαπάνες. Η μόνη ε, περικοπή δαπανών ήταν εις βάρος του κοινωνικού κράτους. Αποτύχαμε λοιπόν. Για μεγαλύτερη ανάπτυξη αποτύχαμε. Είναι η απόλυτη αποτυχία είναι η διαρκής πολιτική λιτότητας και περικοπών. Τώρα επιτρέπονται τα κράτη-μέλη να μπορούν να μειώσουν το έλλειμμα και τις, ε, ε, την υπερχρέωση. Εμείς πρέπει να πούμε ότι εσείς υποβάλλετε τώρα στους λογαριασμούς που έχουν καταστραφεί τα κράτη-μέλη δεν έχουν ούτε μια δεκάρα να επενδύσουν και βλέπουμε ότι τα προβλήματα συνεχίζουν να υφίστανται. Για ποια πράγματα μιλάμε κύριε Επίτροπε, οποιαδήποτε αξιολόγηση πρέπει να είναι σοβαρή και πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα και όχι κάποιους αφηρημένους γενικόλογους στόχους. Οι περικοπές, η λιτότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτά είναι τα αποτελέσματα αυτής της αποτυχίας. Λοιπόν, πρέπει να διαγραφούν αυτά, να είναι, πεταχτούν στα σκουπίδια. Είναι σκουπίδια, αποτυχία απόλυτη. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Ούρτασον έχει το λόγο για τέσσερα λεπτά. Λέει η Ευρωπαϊκή, Επιτροπή, τα ότι τα πρώτα έτη ήταν σχετικά επιτυχή και δείχνουν λέει ότι η μεταρρύθμιση των δημοσιονομικών κανόνων ε, διαδραμάτισε ρόλο σε αυτή την επιτυχία. Ειλικρινά δεν μπορούμε καθόλου να συμμεριστούμε αυτή την άποψη εμείς. Είναι κατεπήγον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μεταθέσει αυτό το στενό εύρος από τη μεχανιστική μείωση των ελλημάτων σε ένα διαφορετικό τρόπο επικέντρωσης. Βλέπουμε ότι η χρέωση, ιδιωτική και δημόσια σε σχέση με τα συστήματα κοινωνικής ε, περίθαψης είχε δραματικές ε, κοινωνικές επιπτώσεις ε, και είχε αποτελέσματα επιζήμια για την ανάκαμψη. Αν αυξήθηκαν αυτά τα επίπεδα χρέωσης και ελλημάτων αντί να μειωθούν. Βλέπουμε λοιπόν όχι μόνο αυτοί οι κανόνες δεν εξυπηρετούν το στόχο αλλά δημιουργούν προβλήματα στην Ευρώπη για μεγαλύτερη ύφεση που προκαλείται. Χρειαζόμαστε μια αντιμετώπιση της κυκλικής αυτής εξέλιξης. Οι κανόνες δεν μπορούν καθόλου αποτελεσματικά να εφαρμοστούν όπως είχαν σχεδιαστεί έχουμε μια ε, διακριτική εφαρμογή τους αντί να χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά. Μετά την οικονομική όμως και ε, κοινωνική ζημιά που προκλήθηκε και είναι κοντόθωρη πολιτική από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λέει ότι δεν υπάρχει ανάγκη να αναθεωρηθούν οι μακροοικονομικές ε, ανισότητες όσον αφορά την επιβάρηση των υπερχρεωμένων χωρών. Χρειαζόμαστε μια πιο συστημική προσέγγιση. Γι' αυτό οι πράσινοι έχουν απογοητευτεί επειδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντιμετωπίζει το πλαίσιο αυτό της οικονομικής διακυβέρνησης ως επιτυχές και λέει ότι δεν χρειάζεται αναθεώρηση. Εμείς όμως πιστεύουμε ότι για να μπορέσει να αντιμετωπιστεί αυτή η κυκλική εμφάνιση αυτών των ε, φαινομένων χρειάζεται μια κωδικοποίηση με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να δημιουργούνται ωφέλη κοινωνικά και περιβαλλοντικά. Πιστεύουμε επίσης ότι πρέπει ιδιαίτερα να αντιμετωπιστούν τα χρέη όσον αφορά την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών Επίτροπε, το μέσο επίπεδο είναι 19% του ΑΕΠ στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το χρέος. Όμως προέρχονται από μέτρα τα οποία παρέχονται στον τραπεζικό τομέα από πλευράς των κρατών μελών. Αυτό δεν μπορεί να θεωρηθεί δίκαιο και πρέπει άμεσα να αντιμετωπιστεί και να αναθεωρηθεί. Χρειαζόμαστε επίσης κωδικοποίηση νομοθετικά κάποιων προσεγγίσεων όσον αφορά τα, τα θέματα τα οποία είναι διαρθωτικού χαρακτήρα. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν αφήσει κανόνες και κανονισμοί γι' αυτό. Στην Ισπανία για παράδειγμα έχουμε εκτίμηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που έχουν, ε, συνεπάγεται ανεργία 20%. Αυτό όμως ε, βλέπουμε ότι δεν αντανακλά πραγματικά ωφέλη για την οικονομία. Χρειάζεται μια αναθεώρηση της προσέγγισης αυτής σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Επίτροπε, είμαστε επίση υπέρ του να ολοκληρωθεί ο πίνακας επιδόσεων για τι ανισότητες με κοινωνικούς δείκτε. Πρέπει να συμπεριληφθούν αυτοί οι κοινωνικοί δείκτε σε αυτήν την αναθεώρηση. Θα θέλαμε να υλοποιηθεί αυτό όπως είχε δηλωθεί. Η εφαρμογή των κανονισμών. Πρέπει να πούμε ότι πρόσφατα τι τελευταίε ημέρε ζητήθηκε από την Επιτροπή από την Ισπανία να συνεχίσει να μειώνει το έλλειμμά τη. Όμως ε, πλήττεται η χώρα αυτή από τεράστιο ποσοστό ανέργων, ανεργίας και αυτοί οι άνεργοι δεν εποφελούνται από κάποια ειδικά κοινωνικά μέτρα. Τι θα έπρεπε να γίνει. Αυτό αν συνεχιστεί ως κατάσταση είναι κοινωνικά τυφλό και αποτελεί αυτοχειρία. Γι' αυτό πιστεύουμε ότι μια αναθεώρηση χρειάζεται κατεπηγόντως ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την στασιμότητα. Ευχαριστώ. Ε, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα τον λόγο έχει ο Στίβεν Γουλφ για το EFTD. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κύριε Ντομπρόφσκης. Περίμενα στην ομιλία σας να παρουσιάσετε με δοξασμένη ιστορία στον αφορά τις δίπτυχες και εξάπτυχες ρυθμίσεις. Πώς βοήθησαν να βγει η Ευρώπη από την ύφεση. Και για μία ακόμη φορά ε, τελικά πετύχατε το στόχο. Χριστούγεννα είναι, μέλη του Κοινοβουλίου. Και είναι Χριστούγεννα που οι γονείς λένε στα παιδιά τους πολλά παραμύθια παραμύθια για το καλό που υπάρχει στον κόσμο όταν γνωρίζουμε ότι υπάρχει κακό εκεί έξω. Και σε αυτή την αίθουσα για μία ακόμη φορά μας είπατε πολλά παραμύθια. Διότι όπως ακούσατε από τα μέλη στο Κοινοβούλιο, το βασικό θέμα των εξάπτυχων ρυθμίσεων είναι ο έλεγχο. Έλεγχο των κυβερνήσεων, των προπολογισμών των κυβερνήσεων, έλεγχο των δαπανών που κυσπούν τι αποφάσει, έλεγχο των λαών τη Ευρώπη, έλεγχο των δημοκρατικά εκλεγμένων κυβερνήσεων, μείωση σταθερότητα, αύξηση του χρέου, μόνο φτώχεια σε όλη την Ευρώπη και τα Χριστούγεννα αυτός ο έλεγχος και η ιστορία των Χριστουγέννων πρέπει να σας δείχνουν γιατί η Ευρώπη ακολουθεί λάθος πορεία. Εκατομμύρια Ευρωπαίοι θα γιορτάζουν τα Χριστούγεννα λέγοντας τα παιδιά τους ότι ο Άι Βασίλης θα τους δίνει δώρα, θα τους φέρει δώρα. Και αν έλεγχε τον Άι Βασίλη η Ευρωπαϊκή Ένωση, η ιστορία θα ήταν διαφορετική. Πρώτα απ' όλα, ο Άι Βασίλης δεν θα μπορούσε να οδηγήσει πάνω από 4,5 ώρες χωρίς να κάνει διάλειμμα 45 λεπτών σύμφωνα με τις οδηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ίσως ακόμα και τα, η τάρανδή του, ο τάρανδός του, ο Λούντολφ θα είχε ταχογράφο. Σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ενώσης θα έπρεπε να έχει και σφραγίδα ε, στο πίσω μέρος του ο τάρανδος με τις σφραγίδες της Ευρωπαϊκής Ενώσης. Και για τις οδηγίες για τα ζώα δεν θα μπορούσε η Βασίλισσα να χρησιμοποιεί καν τον τάρανδο. Και θα, αν δεν υπήρχε οδηγία θα λέγανε τα μέλη ότι πρέπει να δημιουργηθεί ομάδα για να αποφευχθεί η κατάχρηση των ζώων, των ταράνδων του Άι Βασίλη. Και οι επιθεωρητέ Ευρωπαϊκή Ένωση θα ρωτούσαν τον Άι Βασίλη αν συμμορφώθηκε με του κανονισμού. Όπω θα κατέστρεψε η Ευρωπαϊκή Ένωση τον Άι Βασίλη, εσεί καταστρέψατε την ιστορία των Χριστουγέννων, την ίδια για εκατομμύρια Ευρωπαίου, τι οικογένειέ του και για τα παιδιά του. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Μόνο έχει τον λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, μετά την εφαρμογή από την Ένωση του Συμφώνου Σταθερότητα τη Ένωση, ποια είναι η αποτελεσματικότητα τη οικονομική διακυβέρνηση. Οι Γάλλοι πατριώτε διαπιστώνουν το ίδιο με εσά και καταδικάζουν το χρέο στο Αβυσαλέο λόγω τη ιδιωτικοποίηση του δημοσίου χρήματο από τι παγκόσμιε αγορέ κεφαλαίων. Αυτή η υπερχρέωση κάνει σκλάβου του πολίτε του χρέου στο μέλλον. Οι πιστωτέ απαιτούν από εμά περισσότερη λιτότητα συνεχώ. Κοινωνικέ ιδιωτικοποίησει, λιγότερε δημόσιε υπηρεσίε, λιγότερη κυριαρχία όσον αφορά το, το χρέο. Είναι τραγωδία οικονομική και κοινωνική που δημιουργήσατε στην Ελλάδα και στην Κύπρο με τι δικέ σα αλλαγέ. Κάθε κάτω μέλο μπορεί να, αν ήταν ελεύθερο, μπορούσε να μειώνει το έλλειμμά του και το δημόσιο χρέο του, αλλά οι οικονομικέ ε, προσπάθειε ε, πρέπει να αφορούν τι κακέ δαπάνε. Υπερβολικό κόστο τη μαζική μετανάστευση ε, τη συνεχή διάσωση του ευρώ. 17 δισεκατομμύρια το χρόνο επί 4 χρόνια στη Γαλλία. Το κόστο του κοινωνικού ταμείου. Λοιπόν, χωρί λιτότητα πρέπει να επανέλθει η ισορροπία στου υπολογισμού. Χρειάζονται εθνικά μέσα. Έλεγχο των συνόρων, των νομίσματων, των προπολογισμών, των τραπεζών και των εθνικών προτεραιοτήτων. Που η, η φεντεραλιστική σα Ευρώπη τα έχει κατασχέσει όλα αυτά. Εγκαταλείποντα το φανταστικό σα κόσμο και, και, και χάρη σε πατριωτικό οικονομικό μοντέλο θα, θα βρει η Ευρώπη ε, υγιή οικονομικά με ανάπτυξη και απασχόληση. Δεν χρειάζεται το Ηνωμένο Βασίλειο των Six Pack και των ε, Twin Packs για να έχει μικρότερο, μικρότερο χρέο από τη Γαλλία και οικονομική ανάπτυξη πάνω από το 3% φέτο. Ο κύριο Γιούνκερ ε, προσπάθησε να εφαρμόσει δημοσιονομική ε, λιτότητα για να μειώσει το χρέος των άλλων. Λοιπόν, 20% είναι το χρέος όσον αφορά το ΕΠ στην Ευρώπη. Ρωτήστε τον κύριο Αρτούι τι πιστεύει για αυτά που συμβαίνουν στην Γαλλία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και έτσι ολοκληρώνεται αυτός ο γύρος παρεμβάσεων. Περνάμε στις επιμέρους παρεμβάσεις ευρωβουλευτών. Έχετε τον λόγο εσείς. Ε. Ευχαριστώ και ευχαριστώ και τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αυτά τα οποία μας ε, είπε. Πράγματι ασκήθηκε κριτική για το ότι το κείμενο αυτό είναι σύντομο και περιέχει ε, μόνο τα γεγονότα. Εγώ θα ήθελα να σας ε, συγχαρώ και εγώ θα έλεγα πως ε, αν δεν είναι κάτι χαλασμένο δεν ανάγκη να το φτιάξουμε όσον αφορά δηλαδή το Σύμφωνο Σταθερότητας και θεωρώ πως ακριβώς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει ακριβώς να αντιληφθεί ότι πρέπει να εφαρμόσουμε αυτά τα οποία έχουμε συμφωνήσει. Αυτά τα οποία συμφωνήσαμε, αν υπήρχαν και πιο πριν, όπως παραδείγματο χάρη ο μηχανισμός των ανισορροπιών, θα είχαμε αποφύγει δραματικές καταστάσεις που είδαμε σε έναν αριθμό κρατών μελών. Αλλά αυτό το οποίο θεωρώ πως είναι το σημαντικότερο είναι το ότι αυτή τη στιγμή συζητάμε ένα κείμενο το οποίο είναι ξεκάθαρο και σαφές, αλλά υπάρχει μια βρετανική παροιμία η οποία λέει η ουσία του πράγματος φαίνεται, όταν, φαίνεται στην πράξη. Εντάξει, ίσως δεν αφορά τους Βρετανούς αυτή η συζήτηση. Στην πράξη λοιπόν βλέπουμε ότι χρειάζεται μια υγιής βάση για το ευρώ. Και ακριβώς φάνηκε το ότι πρέπει να τηρούμε τις υποσχέσεις που έχουμε ε, δώσει. Και αυτό δεν γίνεται, δεν θα αναφέρω τώρα ονόματα, αλλά ξέρουμε ποιο είναι το κράτος το οποίο έχει κάνει τις μεγαλύτερες ε, παραβάσεις αυτά και όπως είπα θα σας κρίνουμε με βάση τις πράξεις σας. Ευχαριστώ. Κυρία Ντελάνγκε, δέχεστε μία μπλε κάρτα. Ναι. Ο κύριος Χρυσόγονος. Οι δύο ομιλητές του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος μας μίλησαν για την ανάγκη να σεβαστούμε τα συμφωνημένα και τους κανόνες της οικονομικής διακυβέρνησης. Φαίνεται ότι τους διαφεύγει όμως πως στο ευρωπαϊκό δίκαιο εκτός από τους κανόνες οικονομικής διακυβέρνησης υπάρχουν και κανόνες περί δικαιωμάτων παραδείγματος χάρη ο χάρτης θεμελιωδών δικαιωμάτων οι οποίοι παραβιάζονται μέσω της υποτιθέμενης εφαρμογής της οικονομικής διακυβέρνησης που αντί να καταλήξει όμως και αυτή στη βιωσιμότητα του χρέους καταλήγει στο να διονγκώνεται διαρκώς περισσότερο το χρέος και να παραβιάζονται διαρκώς περισσότερο τα κοινωνικά δικαιώματα. Σα ρωτάω λοιπόν μπορούμε να θυσιάζουμε τα κοινωνικά δικαιώματα στο βωμό μιας δίθεν δημοσιονομικής εξυγίανσης. δεν ήταν ερώτηση περισσότερο, αλλά ήταν μάλλον ε, δήλωση. Κοιτάξτε, θα σας πω αυτό το οποίο είπε ο κύριος ε, Ντράγκη δεν είναι ότι έχουμε κάποιο φετιχισμό με τους αριθμούς, απλά οι δεσμεύσεις αυτές είναι ακριβώς η βάση και η άγκυρα της εμπιστοσύνης στην οικονομία μας. Εκεί πέρα βασιζόμαστε, αυτό είναι το θεμέλιο. Αλλιώς υπάρχουν πάρα πολύ σοβαρές συνέπειες. Αυτά δεν γίνονται, ή το ένα ή το άλλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Φερέιρα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 η προσαρμογή η ευρωπαϊκή δεν λειτουργήσε. Πέρασαν έξι χρόνια από την έναρξη της κρίσης και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βρίσκεται στα ίδια σημεία σε σχέση με, με, το, τις άλλες περιοχές. Ε, βρίσκεται σε στασιμότητα. Βρίσκονται εκατομμύρια ανέργων. Μία επιβάρυνση δημοσιονομική από την υπερχρέωση που είναι αφόρητη. Και κατά της κρίσης δράση ήταν αποκλειστικά η νομισματική πολιτική. Όμως τα επιτόκια είναι μηδενικά σχεδόν και ακόμα έτσι η οικονομία δεν ανακάμπτει. Σε αυτή την ανησυχητική κατάσταση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι σκέφτεται για την οικονομία το 2015. Προτείνει μια ουδέτερη, αμερόληπτη οικονομική πολιτική χωρίς επέκταση. Ερωτώ, σε μια ζώνη που δεν έχει ισοτιμίες διαφορετικές, που έχει μια νομισματική πολιτική που έχει εξουδετερωθεί από την κρίση, τι θα πρέπει να γίνει επιπλέον ώστε να προτείνει μια αντικυκλική ε, πολιτική η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καλωσορίζουμε τις προτάσεις της Επιτροπής ε, Juncker. Όμως ε, θα πρέπει να δούμε εδώ την ε, έλλειψη οικονομικής, οικονομικών κινήτρων. Αυτή τη στιγμή σε σχέση με τα six pack αυτά που βλέπουμε ότι νομοθετική, νομοθετικά η προσαρμογή σε τρεις όρους πρέπει να αντιμετωπιστεί. Για αν υπάρχει εξωτερική, εξωτερικό πλήγμα σε σχέση με τα κράτη μελη και διαφθορτικά μέτρα που θα πρέπει να υιοθετηθούν για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Όμως οι αυθεντικές μεταρρυθμίσεις ε, θα πρέπει να εξεταστούν. Ε, ερωτώ, ποια μέτρα θα υιοθετήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχει κάτι υπόψη, όχι. Όλοι, όλες οι προσαρμογές στο χρονοδιάγραμμα σε σχέση με τα δημοσιονομικά παρουσιάστηκαν ως πολιτικά μέτρα σε μια πολιτική προσέγγιση. Είναι όμως ε, ακριβώς αυτό το οποίο πρέπει να επικεντρωθούμε να αλλάξει η ημερήσια διάταξη. Διότι αν δεν υπάρξει κάποια αλλαγή στην πολιτική αντιμετώπιση ανεργίας δεν θα υπάρξουν ισορροπημένα δημοσιονομικά. Πρέπει να δούμε την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Αρνείται η Ευρώπη να το κάνει και αυτή τη στιγμή προκαλούμε μια κατάσταση που δεν είναι αποτελεσματική. Να αλλάξει η ημερήσια διάταξη παρακαλούμε. Ευχαριστώ. Ε, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, κύριε Σάντα, παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Δεν είναι εύκολο βεβαίως το να κρίνει κανείς τους διαφόρους προϋπολογισμούς και βλέπουμε τώρα τι γίνεται στο Βέλγιο που για πρώτη φορά μετά από 25 χρόνια προσπαθεί μια κυβέρνηση να περιορίσει τις δαπάνες και για πρώτη φορά δεν έχουμε αύξηση των δαπανών αλλά πάμε προς μια εξυγίανση. Όμως είναι αναγκαία ε, μια τέτοια κίνηση αν θέλουμε να βοηθήσουμε την ανάπτυξη και τις ε, δουλειές. Ε, αλλιώς βλέπουμε πως δεν υπάρχει καμία εμπιστοσύνη για το μέλλον. Ε, βεβαίως βλέπουμε τις πάρα πολλές απεργίες που υπάρχουν. Αλλά η εμπιστοσύνη είναι λέξη κλειδί. Χωρίς εμπιστοσύνη δεν υπάρχουν επενδύσεις, δεν υπάρχει ανάπτυξη, δεν υπάρχουν δουλειές. Αλλά η εμπιστοσύνη αυτή θα έρθει μόνο εάν τηρήσουμε σταθερή την πορεία σε αυτά τα οποία έχουν συμφωνηθεί. Και το επενδυτικό το σχέδιο των 300 δισεκατομμυρίων μπορεί να ακούγεται καλό, αλλά τα λεφτά θα πάνε πεταμένα εάν δεν κάνουμε τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις. Γι' αυτό ακριβώς φοβάμαι πως ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι υπερβολικά θετική στην αξιολόγηση για το διπλό και το εξαπλό πακέτο. Ναι, λήψει πράγματι, αλλά ταυτόχρονα ε, έχει αυξηθεί το χρέος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι το οποίο υποσκάπτει την απαραίτητη, όπως είπα, εμπιστοσύνη. χαλάρωση είναι μια πολυτέλεια που δεν την έχουμε αυτή τη ε, στιγμή. Πρέπει να διατηρήσουμε σταθερή την πορεία για να διατηρήσουμε, όπως σας είπα, ε, την απαραίτητη εμπιστοσύνη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Τόιρερ έχει το λόγο για ένα λεπτό και 30 δευτερόλεπτα. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, η υπερχρέωση των κρατών κατά μέσο όρο πριν από την εισαγωγή του ευρώ ήταν υπερβολικά υψηλή και πριν από την κρίση την οικονομική και δημοσιονομική ήταν υπερβολικά υψηλή και εξακολουθεί να είναι υψηλή. Γι' αυτό είναι αξιοπερίεργο ότι κάποιοι συνάδελφοι ζητούν να συνεχίσει η χρέωση ώστε να αντιμετωπιστεί η υπερχρέωση του παρελθόντος. Δεν είναι η σωστή πορεία αυτή. Πρέπει να αποφύγουμε την παγίδα της υπερχρέωσης και αυτό γίνεται μόνο με διαφορετικές μεταρρυθμίσεις. Πρέπει θεσμικά να μπορέσει να επιβληθεί το κοινό κοινοτικό συμφέρον. Και αυτό έγινε με τα εξαπλά και τα διπλά μέτρα για την, ε, το μέτρο ανάπτυξης, ε, για το Σύμφωνο Ανάπτυξης και Σταθερότητας ε, που από την Ομοσπονδιακή Γερμανία και τη Γαλλία παραβιάστηκε ευθύ εξ αρχής. Όποιος δεν τηρεί τις τα συμπεφωνημένα υπονομεύει την πορεία της Ένωσης. Αποφασιστικό είναι οι κανονισμοί να εφαρμόζονται. Και εδώ, Επίτροπε Ντομπρόφσκι, βασιζόμαστε σε εσά με τις ελπίδες μας. Αποδείξατε πως στη Λετωνία μια χώρα με μεταρρυθμίσεις μπορεί να επανέλθει σε μια πορεία ανάκαμψης και ανάπτυξης. Η Ελλάδα, η Πορτογαλία, η Ιρλανδία, η Ισπανία έκαναν μεγάλες προσπάθειες. Έσφιξαν το ζωνάρι οι πολίτες. Βλέπουμε τώρα το φως στην άκρη της σύραγγας. Οι χώρες αυτές επανήλθαν σε μια πορεία ανάπτυξης. Το αποφασιστικό ερώτημα είναι τι θα κάνουν η Γαλλία και η Ιταλία. Και εδώ πρέπει να μεριμνήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι κανονισμοί να εφαρμόζονται από τις μεγάλες χώρες και όχι μόνο από τι μικρές. Από κοινού πρέπει να εφαρμόζονται οι κανόνες. Αυτό αναμένουμε. Ευελπιστούμε Ευχαριστούμε Επίτροπε Ντομπρόφσκης ότι αυτό θα επιβάλλεται με την Επιτροπή. Ευχαριστώ. Ε, Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν έχετε μπλε κάρτα. Κύριε Έθριτζ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Συμφωνείτε μαζί μου ότι αν σκέφτεστε τα εξαπλά ε, ε, πακέτα θυμίζει τον Κριστιανό Ρονάλντο, που είναι κάτι πολύ θετικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση, θυμίζει τους μης. Αλλά τελικά θυμίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι, δείχνει κάτι το οποίο είναι πολύ χαλαρό, πλαδαρό η εικόνα της ε, ε Ευρώπης. Όχι σαν τον Ρονάλντο, είναι σαν εμένα όταν ξυπνάω εγώ το πρωί. Μήπως έτσι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και να παρουσιάσουμε και τη φυσική κατάσταση Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχετε τώρα, είναι ενδιαφέρουσα η ερώτηση, έχετε τον λόγο να απαντήσετε. Ευχαριστώ για τον καθορισμό εξάπτυχο ή εξαπλάν, είναι σωστή διατύπωση. Είναι σαφέ όμω ότι αυτό που προσέχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ότι πολλέ φορέ δεν πιστεύουμε αυτά που κάνουμε. Όταν συζητούμε με ανθρώπου από άλλε περιοχέ, από την Ινδία, από τον χώρο του Ειρηνικού και μα λένε τι κάνετε στην Ευρώπη, έχετε υποδομέ, έχετε εξαιρετικά πανεπιστήμια, εξαιρετικά συστήματα υγειονομική περίθαψη. Αν δεν τα καταφέρετε εσεί να επανέλθετε στη σωστή πορεία, ποιο θα τα καταφέρει. Το ευρώ δεν είναι ούτε αίτιο ούτε η λύση των προβλημάτων. Πρέπει να δούμε στην πραγματική οικονομία, τεχνολογία, καινοτομία, ανάπτυξη. Και τότε πιστεύω ότι μπορούμε με τα εξαπλά όπως ένας ε, αθλητής που έχει προπονηθεί να τα καταφέρουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αντιλαμβάνομαι πως είναι σημαντικό το θέμα και ότι αισθάνεστε και κάποια ευθύνη, αλλά σας παρακαλώ πάρα πολύ μία μπλε κάρτα θα επιτρέψω και όσοι το ζήτησαν αργότερα δυστυχώς δεν θα μπορέσουν να λάβουν το λόγο. Ο κύριος έχει τώρα το λόγο. E για μας είναι σημαντικό για τα εξαπλά και τα διπλά μέτρα. Έχουμε έναν μηχανισμό που δημιουργήθηκε να ευθυγραμμιστούν τα κράτη-μέλη με τα συμφέροντα των μεγάλων επιχειρήσεων που είναι εκείνες που διακυβερνούν την Ευρώπη. Και βλέπουμε ότι υπάρχει η ανάγκη αυτής της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και υιοθετείται μια νομισματική ε, πολιτική λιτότητας που εξυπηρετεί, πάντα τα ίδια συμφέροντα. Δημιουργείται λοιπόν μια κατάσταση ανισόρροπη. Υπάρχουν τρία θέματα. Πρώτα, πώς επεξηγείται ότι σε σχέση με τα κράτη-μέλη ε, βρίσκουμε ότι παραβιάζουν τα κράτη αυτούς τους κανόνες που θεωρούμε ότι είναι απόλυτα ανεπαρκείς. Δεύτερον, λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι υπάρχουν πρόοδοι ότι το χρέος και το έλλειμμα μειώνονται. Αν συμβαίνει αυτό, γιατί συνεχίζουμε να βρισκόμαστε στην κρίση χωρίς προοπτικές. Τρίτον, πώς επεξηγείται το ότι κατά τη διάρκεια αυτής της κρίσης τα κράτη-μέλη εκτός ευρώ ε, είχαν μεγαλύτερη ανάπτυξη σε σχέση με τα κράτη ευρώ. Ή τα κράτη που αποφάσισαν να διατηρήσουν την νομισματική κυριαρχία τους έχουν μεγαλύτερη ανάπτυξη. Πώς το εξηγείτε. Ευχαριστώ Σβέν Γκίγκολτ ε, έχει το λόγο. Κύριε, Κύριε Επίτροπε, έχετε μια επανεξέταση που γίνεται εδώ των κανόνων και κανονισμών που αναθεωρήθηκαν. Ήταν ένα πίμαχο θέμα νομοθετικό αυτών των προτάσεων. Στην επανεξέταση η κατάσταση αυτή ε, τονίζεται ιδιαίτερα διότι οι κανονισμοί που εδώ εγκρίναμε δεν έχουν τέτοια μορφή ώστε πραγματικά να εφαρμόζονται αποτελεσματικά και να δημιουργούν και κάποια διαφάνεια για το αν αυτοί οι κανονισμοί εφαρμόζονται πραγματικά. Αν δούμε το τι συμβαίνει, τα διαθωτικά ελλείμματα των κρατών μελών μειώθηκαν όπως είχε συμφωνηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Από 18 κράτη 14 τα μέτρα τα οποία είχαν συμφωνηθεί από 14 κράτη δεν υλοποιήθηκαν. Από κάποιους συναδέλφους τώρα ακούμε ότι δεν υπάρχουν λέει προβλήματα πρέπει να εφαρμοστούν αυστηρά αυτοί οι κανονισμοί. Αν γινόταν αυτό όμως ε, τότε η Ευρώπη θα υπαναχωρούσε σε ένα επίπεδο ύφεση. Πρέπει να δημιουργηθεί μια δυνατότητα να ανακάμψουμε. Δεν μπορεί να λέει κανείς οι κανόνες και οι κανονισμοί αυτοί είναι εξαιρετικοί. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν συνάδελφοι που λένε ότι αυτούς τους πιο περίπλοκους κανόνες πρέπει να τους καταστήσουμε πιο εύληπτους και απλούς. Όμως η κατάσταση είναι προκυκλή Γι' αυτό η απάντηση στα προβλήματα σε σχέση με τους πιο αυστηρούς κανόνες του Συμφώνου Ανάπτυξης και ε, ε, ε, Οικονομικών Επενδύσεων είναι μια πολιτική που θα οδηγήσει σε προσαρμογές. Χρειάζεται τα κράτη τα οποία είναι ισχυρότερα οικονομικά να επενδύσουν περισσότερα ώστε να υπάρξει μεγαλύτερο περιθώριο για άλλα κράτη να εξηγιάνουν τα δημοσιονομικά τους. Τι κάνει όμως το Συμβούλιο και τα κράτη-μέλη, τι κάνουν. Δεν υλοποιούν μια τέτοια πολιτική σε σχέση με τον Ντράγκη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας τον αφήνουν μόνο του και δεν τον υποστηρίζουν που προσπαθεί να στηρίξει τα κράτη αυτά. Γι' αυτό λοιπόν Επίτροπε σε σχέση με το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης πορεύεστε προς την ορθή κατεύθυνση. Όμως όλα αυτά τα προβλήματα που υπάρχουν δεν ονοματίζονται, δεν ονομάζονται ε, το ένα με το άλλο με το σωστό τρόπο. Και το Συμβούλιο δεν είναι πρόθυμο να αναλάβει τις ευθύνες του για την πολιτική που χρειάζεται η Ευρώπη. Ευχαριστώ. You have a blue card. Έχετε μια μπλε κάρτα κύριε Γκίγκολτ. Τη δεχόσαστε ως ερώτηση. Ευχαριστώ. Φυσικά. Έχετε τον λόγο εσεί, κύριε Λουκάς. Κύριε Γκούγκερ, κύριε Γκίγκολτ, είπατε οι απλοί κανόνες είναι προκυκλικοί, είπατε. Αν έχουμε ένα κράτος το οποίο έχει ισοσκελισμένο προϋπολογισμό, με τους απλούς κανόνες ε, η υπερχρέωση μπορεί να φτάσει στο 3%. Σε ένα κράτος με 20% τι σημαίνει αυτό, ότι κατά 15% θα μπορέσουν να επεκταθούν οι δημόσιες δαπάνες. Τι είναι προκυκλικό εδώ, για τη δυνατότητα που εσείς επισημάνατε με αυτή την εφαρμογή. Ευχαριστώ. Ακούστε, το πρόβλημα δεν ήταν ότι η κατάσταση ε, λειτουργούσε ή όχι. Πράγματι, τα κράτη της Ευρωζώνης ε, αυτόν τον κανόνα του 3% τον ε, τηρούσαν ή τον ξεπερνούσαν. Το πρόβλημα ήταν ότι δεν είχαμε κανόνες να μεριμνούμε το επίπεδο υπερχρέωσης να μειώνεται πάλι ξανά. Κατά τούτο λοιπόν οι παλαιοί κανόνες για το 3% ή 60% ήταν λοιπόν πρωτό, λύσεις εξαπλουστευτικές δεν έδιναν λύσεις στο πρόβλημα. Και γι' αυτό ειλικρινά τα όσα είπατε εσείς είναι υπεραπλουστευτικά και ε, η επικέντρωση μόνο στην αρνητική φάση είναι μονομερής, μονόπλευρη. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Μάρκο Βάλλη έχει το λόγο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, κοιτάξτε μας σας παρακαλώ. Κύριε Επίτροπε, τίποτα. Σε αυτή τη φάση μιλώνω ονόματι του 21% των Ιταλών που πήγαν να ψηφίσουν στις τελευταίες ευρωεκλογέ. Αυτά τα άνομα καταπιεσμένα από την κρίση έδωσαν την ψήφο σε μένα για να έρθω εδώ και να σα πω ότι εμεί δεν θέλουμε πλέον το σύμφωνο σταθερότητα. Δεν θέλουμε πλέον δεσμού για του προπολογισμού. Δεν θέλουμε πλέον να είναι οι λογιστέ τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για λογαριασμό των, ε, των αγορών να ρυθμίζουν τα δημοσιονομικά των μελών. Θέλουμε πολιτικού που να βλέπουν το υπερβολικό σπρέτ, την κερδοσκοπία, ε, τις, κερδοσκοπικέ επιχειρήσει των τραπεζών. Αλλά εμεί να θεσπίζουμε του κανόνε και όχι εσεί. Ε, η ευημερία των περισσότερων πολιτών με αυτέ τι επιβολέ φορολογικέ έρχεται μετά από τα συμφέροντα των κερδοσκόπων και αυτό δεν μπορούμε να το δεχτούμε. Το σύμφωνο σταθερότητα και ανάπτυξη είναι κάτι τοπικό. Η σταθερότητα στι χώρε με μεγάλο χρέο είδαμε οδηγεί μόνο στη φτώχεια, στην ανεργία και ξεπολύει ε, την ιδιοκτησία των κρατών μελών ε, και δημιουργείται προς την αγορά που είναι κάτι αφηρημένο και εξυπηρετεί τα συμφέροντα των 1% του πληθυσμού. Λοιπόν, δεν πιστεύει πλέον ο λαό στην πολιτική. Οι περισσότεροι δεν πάνε να ψηφίσουν και ζουν σε ένα σύστημα ε, που απεχθάνονται. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε σωστό και δίκαιο με το σύμφωνο σταθερότητα, με το εξαπλό και διπλό σύμφωνο είναι αυτό βλέποντας ότι εσείς δεν έχετε την ηθική και διανοητική ειλικρίνεια να το κάνετε όπως ε, αλλού. Και έχει, ε, ε, όπως είδαμε και τον Λουξ Λίξ και πέρασε ο κόσμος, καλούμε να, στο δημοψήφισμα στην Ιταλία για το ευρώ. Και εκεί θα φέσουν οι μάσκες όσον αφορά την δικτατορία, την οικονομική επιβάλληση στις δημοκρατίες. Θα πρέπει να δούμε ποιος φταίει πραγματικά για την κρίση, ποιος έφερε τη χώρα μας στο ενιαίο νόμισμα καλύπτοντας τους λογαριασμούς και ποιος έκλειψε τα δημοσιονομικά και από την κυριαρχία των λαών. Το, και από και τα πούλησε στην αγορά και οι ιδιωτικέ τράπεζες κερδοσκοπούν. Κοιτάξτε με στα μάτια όταν εγώ σας μιλώ. Εμείς εκπροσωπούμε εκείνους που δεν θα παραιτηθούν ποτέ, δεν θα είναι ε, πλέον δούλοι του χρέους και της τεχνοκρατίας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Βαλή. Χρησιμοποίησατε κάποια σκληρά λόγια. Καλό είναι να το ξανασκεφτείτε, να τα ξανασκεφτείτε πριν την επόμενη παρέμβασή σας. Και α, σας ακούει ο Επίτροπος ακόμα και αν δεν σας βλέπει. Λοιπόν, ο κύριος Ζαριανόπουλος τώρα έχει το λόγο. Για ένα μισή λεπτό. Μεγαλύτερους και ισχυρότερους. Μεγαλύτερη μόνιμη ανεργία και φτώχεια για περισσότερους. Με εργαλεία το σύμφωνο σταθερότητας, τα ευρωπαϊκά εξάμεινα, τα δίπτυχα και εξάπτυχα μέτρων τη στρατηγική. 2020. Δεν είναι λάθος ούτε πρόσκαιρη ανάγκη. Είναι ο λόγος ύπαρξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χρειάζεται την ανεργία και την ευέλικτη εργασία για πάφθηνους μισθούς. Μισθούς ψίχουλα για τα κέρδη που επιδοτείται με νέα κεφάλαια, άγριους φόρους, κλοπή και κατεδάφιση της κοινωνικής ασφάλισης. Χρειάζεστε κέρδη για ανταγωνιστικότητα γιατί χωρίς αυτή δεν υπάρχει αναθεωρείται τη λεγόμενη οικονομική διακυβέρνηση για πιο γρήγορη και αποτελεσματική επιβολή αντιλαϊκών μέτρων σιδερένια εποπτεία και πειθαρχία μνημόνια διαρκείας για όλα τα κράτη. σφίγγεται τη θηλιά στους λαούς για να κινηθεί η οικονομική μηχανή που ακόμα δεν παίρνει μπρος παρά τις λαϊκές θυσίες και τα δισεκατομμύρια που την ταΐζετε. η κρίση είναι στη μήτρα του συστήματός σας. εσείς το ξέρετε ότι δεν αλλάζετε και όσοι λένε ότι θα σας μεταμορφώσουν από σφαγείο σε παράδεισο λένε ξεδιάντροπα ψέματα. οι λαοί πρέπει να μάθουν. Αυτή είναι ισχυρή και όχι τα μονοπόλια η ευρωπαϊκή ένωση οι κυβερνήσεις και τα κόμματά της που κάθονται στο σβέρκο τους. ούτε φόβος λοιπόν ούτε αναμονή. πριν τους πάρουν και την τελευταία βουκιά επίθεση τώρα για διέξοδο που να υπηρετεί τα λαϊκά συμφέροντα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Λαμασούρ έχει το λόγο για δύο λεπτά, παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αυτά που είπατε το επιβεβαιώνουν κύριε την της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το πρόβλημα δεν είναι αναθεώρηση των κανόνων που θεσπίστηκαν στην ακμή του, ε, της κρίσεως για να εξηγενθούν τα δημοσιονομικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται πραγματικά περί εφαρμογής των κανόνων αυτών και να εφαρμοστούν πλήρως στο γράμμα και στο πνεύμα. Είναι ένα θέμα αξιοπιστίας αξιοπιστίας της Ενώσεως και πιο συγκεκριμένα της διακυβερνήσεως της Ευρωζώνης που έχει πρικοδοτηθεί με στόχους έτη περαιτέρω φιλοδόξου στον τομέα αυτό με τη συνθήκη που λέγεται ε, Οικονομικό Σύμφωνο, το Fiscal Compact και αφορά και την αξιοπιστία της Νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και μετά τους συναδέλφους του ΕΛΚ και κυρίω του κυρίου Τόιρερ θα ήθελα και εγώ να κάνω μια προειδοποίηση. Οι κανόνε θα πρέπει να εφαρμόζονται ταυτόσημα σε όλες τις χώρες ανεξάρτητα από το μέγεθος αυτών. Υπενθυμίζω ότι αν έπρεπε να θετηθεί μια νέα νομοθεσία Six Pack και Twin Pack είναι διότι οι αρχικοί κανόνε το Σύμφωνο σταθερότητα και ανάπτυξη, ε, δεν εφαρμόστηκαν. Ε, το 2003 Είδαμε ότι οι δύο μεγαλύτερες οικονομικές δυνάμεις της Ενώσεως, η Γερμανία και η Γαλλία, βγήκαν ε, ταυτόχρονα ε, από τα όρια. Ζήτησαν και πέτυχαν χωρίς δυσκολία μια ευελιξία, μια ερμηνεία των κανόνων ε, που έθεσε εν κενό το περιεχόμενο. Και το συμπέρασμα που συναγάγαμε ήταν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορούσε να λειτουργήσει επί τη βάση μιας αρχής κρυφής ε, που, που είναι μεγάλες χώρες που δεν είναι πολύ μεγάλες για να αποτύχουν αλλά πολύ μεγάλες για να τιμωρηθούν ή να κατηγορηθούν. Αν ξαναρχίσουμε σήμερα, αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δείξει ότι είναι άκαμπτη έναντι της Ελλάδας και έναντι της Πορτογαλίας αλλά τρέμει έναντι των χωρών ούτως υπήν μεγαλύτερων της Ισπανίας τότε όλα θα καταρρεύσουν σαν μηχανισμοί διότι τελικά θα ξαναπέσουμε σίγουρα στην κατάσταση που θέλαμε βάσει θυσία να αποφύγουμε. Δηλαδή, εκεί οι χρηματοπιστωτικοί φορείς και οι διάφοροι ε, ε και οι διάφοροι εκείνοι οίκοι βαθμολόγησης θα ασκούν την πολιτική αντί από τους νόμιμα ερετούς εκπροσώπους του λαού. Κύριε Κυρία Λαμασούρ, έχετε γαλάζια κάρτα. Δεχόσαστε να απαντήσετε στην ερώτηση. Έχετε το λόγο. Κύριε Ρόπε. Σας e, e, ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε κάποιες χώρες η κατάσταση είναι διαφορετική βεβαίω. αλλά εγώ θα ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση. Θα πρέπει να υπάρχει κάποια αρχή που θα μας επιτρέπει να υπερασπιζόμαστε τον, ε, τους ανθρώπους μας και ότι όταν θα έχουμε καλύτερα οικονομικά πρέπει να αποκαταστήσουμε το μισθό, το σύστημα κοινωνικής πρόνοιας και τότε μόνο να μιλήσουμε για εφαρμογή νέων προγραμμάτων. Ευχαριστώ. Κύριε Λαμασούρ. Υποθέτεται ότι το πρόβλημα ήδη έχει ρυθμιστεί όταν δυστυχώς μια χώρα κατά διάρκεια σειρά ετών έζησε ε, πάνω από τα μέσα που διαθέτει. Υποχρεώθηκε να ζητήσει από του εταίρου βοήθεια και το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει τότε είναι να αποκαταστήσει την κατάσταση και τα δημοσιονομικά, να τα θέσει εντάξει στη χώρα με τη βοήθεια των εταίρων και μετά μόνο από τη στιγμή που ξεκινήσει ξανά η δημιουργία πλούτου, από εκείνη τη στιγμή μπορεί να γίνει η ανακατανομή της αγοραστικής δύναμης. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Η κυρία Ροντρίγκε τώρα για δύο λεπτά. Κύριε Αντιπρόεδρε, ναι, το νέο πλαίσιο οικονομικής διακυβέρνησης είχε κάποια προβλήματα, έλυσε κάποια προβλήματα, αλλά άλλα δημιούργησε. Η Ευρώπη τώρα είναι παγιδευμένη σε μια στασιμότητα, υψηλή ανεργία, υψηλό, υψηλό χρέος, κίνδυνος αποπληθωρισμού και είναι ε, και διαιρεμένη ε, λόγω των μεγάλων οικονομικών και κοινωνικών αποκλήσεων που γίνονται μετά και πολιτικές αποκλήσεις. Η Κομισιόν αναγνώρισε την κατάσταση στην ε, τελευταία της ε, έκθεση για την ανάπτυξη και τώρα πρέπει να κάνει κάτι για αυτά τα προβλήματα με το να προσαρμόσει το πλαίσιο αυτό οικονομικής διακυβέρνησης. Το πρώτο που πρέπει να γίνει νομίζω είναι να υπάρξει μεγαλύτερο περιθώριο για τις επενδύσεις στο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης και να διασφαλιστεί πως οι συνεισφορές των κρατών μελών στο νέο αυτό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων να είναι ουδέτερες ως προς το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης και δεύτερον χρειαζόμαστε μια πιο ισορροπημένη μακροοικονομική παρακολούθηση που δεν θα κοιτάει μόνο τα οικονομικά αλλά και τα κοινωνικά προβλήματα και τέλος κύριε Αντιπρόεδρε. Ειλικρινά δεν πιστεύω πως υπάρχει πραγματική ε, λύση για τη μείωση αυτών των αποκλήσεων που υπάρχουν στην Ευρωζώνη εάν δεν μπορέσουμε να προωθήσουμε το θέμα αυτό της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης να ολοκληρωθεί δηλαδή η Τραπεζική Ένωση αλλά οπωσδήποτε και να δημιουργηθεί μια πραγματική ε, φορολογική ικανότητα στην Ευρωζώνη. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Ροντρίγκες, έχετε μία μπλε κάρτα. Τη δέχεστε από τον κύριο Κόμπερν. Με ακούτε? Η κυρία Βουλευτής ε, συμφωνεί μαζί μου πως ε, τα ευρωπαϊκά έθνη εκτός του ευρώ τα πάνε σχετικά καλά. Ενώ αυτά εντός του ευρώ δεν τα πάνε καλά. Το ευρώ είναι ένα πολιτικό νόμισμα που δημιούργησε η Κομισιόν για τους δικούς της πολιτικούς στόχους. Και μέχρι να το απορρίψουμε δεν υπάρχει ελπίδα ανάκαμψης για τους λαούς της Νότιας Ευρώπης. Προτείνω λοιπόν στο σώμα η Κομισιόν να παραδεχτεί το λάθος της και να παρατήσει αυτό το νόμισμα. Η κυρία μας το είπε πως είναι προφανές πως αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν, δεν ήταν ακριβώς ε, ερώτηση αλλά δήλωση. Τέλος πάντων. Πράγματι υπάρχει πρόβλημα, αλλά το πρόβλημα δεν είναι το ευρώ. Το ευρώ μπορεί να είναι δύναμη για τα κράτη-μέλη. Το πρόβλημα είναι η οργάνωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης που δεν είναι ισορροπημένη και φαίνεται αυτό τώρα. Γι' αυτό πρέπει να ολοκληρωθεί η Τραπεζική Ένωση για να υπάρχει ένα σωστός οικονομικός συντονισμός μεταξύ ελληματικών και πλεονασματικών χωρών και να υπάρξει όπως σας είπα δημοσιονομική ικανότητα. Αυτό μας λείπει. Σας ευχαριστώ. Τον λόγο τώρα έχει ο κύριος Άσλι ε, Φόξ για ένα μισή λεπτό. Ε, ευχαριστώ Πρόεδρε. Κάθε συζήτηση για την οικονομική διακυβέρνηση με κάνει να είμαι πιο ευγνώμων για το ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν έχει προσχωρήσει στη ζώνη ευρώ. Εγώ πιστεύω ότι είναι βαθιά μη δημοκρατικό για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λέει στα κράτη-μέλη τι θα πρέπει να εισπράττουν και τι θα πρέπει να δαπανούν. Αλλά αυτό είναι η συνέπεια του να εισέρχεται κανείς σε ένα ενιαίο νόμισμα. Και όλο και πιο πολύ γίνεται σαφές ότι το ευρώ ως ενιαίο νόμισμα δεν λειτουργεί. Δεν λειτουργεί για τις πολυισχυδείς οικονομίες ε, στα, που έχει στους κόλπους του. Σαν αποτέλεσμα εκατομμύρια νέων είναι άνεργοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ανεργία των νέων είναι 40% στην Ιταλία, 55% στην Ισπανία, 58% ανεργία των νέων στην Ελλάδα. Τραγωδία για εκατομμύρια οικογενειών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης ε, είναι σωστό το ότι θα πρέπει να, ελέγχεται, να ελέγχονται τα έσοδα και οι δαπάνε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά θα πρέπει να, να συνοδεύεται από τι σωστέ νομισματικέ πολιτικέ. Και αυτό είναι ανέφικτο να επιτευχθεί από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ό,τι και να λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Οικονομική Διακυβέρνηση δεν αναγνωρίζει τα, τα βασικά ελλείμματα και ελλείψεις που υπάρχουν στην οικοδόμηση του ευρώ. Ένα ενιαίο επιτόκιο ποτέ δεν θα είναι σωστό και αποτελεσματικό για όλα τα μέλη της Ευρωπαϊκής Νομισματικής Ένωσης. Και κύριε Ντομπρόφσκης, αν θέλετε να ανθίσει η Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση, τότε τα θέματα των ε, φορολογικών μεταφορών ε, δεν θα πρέπει να εξεταστούν των δημοσιονομικών μεταφορών σε σχέση με τον καθορισμό ενός ενιαίου επιτοκίου. Να λέτε μετά στις κυβερνήσεις της Ιταλίας και της Ελλάδας τι θα πρέπει να γίνεται χωρίς να μεταφέρετε κονδύλια από τα πλουσιότερα μέλη στα φτωχότερα μέλη. Και αυτό είναι κάτι που δεν θέλετε να κάνετε γιατί φοβόσαστε να το πράξετε. Ε, Έχετε μια μπλε κάρτα από ε, συνάδελφο. Την δέχεστε. Ευχαριστώ. Έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Φόξ. Μπορώ να δεχτώ το ότι επικρίνεται και κάνετε επικρίσεις, δεν καταλαβαίνω όμως την αντίφαση που θέσατε. Διότι είπατε ότι υπάρχει ανάγκη νομισματική ένωση, δεν χρειάζεται νομισματική ένωση, αλλά ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποια είναι η λύση. Είναι εύκολο να επικρίνετε. Δεν προτείνετε όμως λύσεις. Από την αρχή της συνεδριάσεως η ομάδα σας επικρίνει. Είστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειαζόμαστε μια νομισματική ένωση για σωστή διακυβέρνηση. Αλλά προτείνετε κι εσείς κάτι. Well, I think that... Νομίζω ότι η Νομισματική Ένωση μεταξύ μικρού αριθμού κρατών μελών που έχουν συγκλίνουσες οικονομίες, παράδειγμα Γερμανία, Ολλανδία, Αυστρία, Φινλανδία, θα μπορούσε να είχε στεφθεί με επιτυχία μια τέτοια νομισματική ένωση. Το πρόβλημα όμως ήταν το ευρώ ήταν πολιτικό εγχείρημα, αντιοικονομικό εγχείρημα. Αν θέλουμε να λειτουργήσει, τότε είτε θα πρέπει με οργανωμένο, διοργανωμένο τρόπο αυτά τα κρέτη που δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε σχέση με την Ελλάδα και την Κύπρο να μπορέσουν να αποχωρήσουν με διοργανωμένο τρόπο. Ή διαφορετικά τα πλουσιότερα κράτη θα πρέπει να πληρώνουν σε αυτά τα ανεπαρκή κράτη-μέλη τεράστια κονδύλια, όπως ε, γίνεται μεταξύ πολιτιών στη ΣΥΠΑ. Ένα από τα δύο θα πρέπει να γίνεται, αλλά δεν συζητείται αυτό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε, κύριε Φόξ. Και στη συνέχεια έχει 1,5 λεπτό τρεμόσα η Μπαρσέλ. Σε ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητέ επίτροπε, είναι πολύ νωρί να κρίνει κανεί αν τα εξάπτυχα και δίπτυχα μέτρα πρέπει να αναθεωρηθούν. Πρέπει να υπενθυμίσω ότι μόλι πριν δύο χρόνια, όταν διαπραγματευόμασταν τα θέματα αυτά του δίπτυχου, της δίπτυχης πρότασης, εμείς πιστεύουμε ότι για μία αναθεώρηση πρέπει να δούμε πώς θα υπολογίζεται το δημόσιο χρέο. Θα συνυπολογίζεται σε αυτό το χρέο των δημοσίων κρατικών υπηρεσιών. Νομίζω ναι και αυτό θα είναι μία από τις ε, μελλοντικέ ιδέες μας για τις μελλοντικέ συζητήσεις για αυτό το θέμα. Για την αναθεώρηση της οικονομικής διακυβέρνησης στην Ευρώπη πρέπει να εξετάσουμε επίσης και τις περιφερειακές ε, και τοπικές κυβερνήσεις με νομοθετικές αρμοδιότητες. Αυτές οι αρχές πρέπει σε σχέση με τις ε, δαπάνες τους ε, να βρίσκονται σε αναλογία με τα έσοδα. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να διασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρχει διαφορετική μεταχείριση διαφορετικών επιπέδων διακυβέρνησης. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για χώρες όπου οι κοινωνικές δαπάνες, οι περισσότερες από αυτές γίνονται σε περιφερειακό επίπεδο. Όμως τα έσοδα φορολογικά και άλλα βρίσκονται επικεντρωμένα στην κεντρική κυβέρνηση. Έχω την εντύπωση ότι θα πρέπει να δούμε περισσότερο το πρότυπο των υπ ΣΥΠΑ, συνάδελφοι. Τι δηλαδή έκανε η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση στη ΣΥΠΑ, πώς δημιουργήθηκε και πώς δημιούργησαν αυτή την Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Διερωτώ με, η πρόταση bailout δεν θα έπρεπε να αναλυθεί για τη μελλοντική μας διακυβέρνηση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Τραμόσα. Και τώρα ο κύριος Λόπετ Μπερμέχο παρακαλώ έχει τον λόγο κυρία Λόπε Μπερμέχο άρχισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την έλλειψη των, ε, ε, του σεβασμού κανονισμών να κατηγορεί τα κράτη-μέλη. Ξέχασε τα κράτη-μέλη που, που δεν τηρούσαν αυτές τις ε, διατάξεις μεταξύ αυτών ήταν η Γερμανία. Και βλέπουμε ότι με μια επισφαλή αγορά εργασίας η Ισπανία που προσπαθούσε να τηρήσει αυτές τις διατάξεις σήμερα έχουμε 25% ανεργία στην Ισπανία και έχουμε το δεύτερο υψηλότερο, την δεύτερη υψηλότερη υπερχρέωση παγκόσμια. Και τι γίνεται με τη διακυβέρνηση. Δεν μπορεί παρά η αξιολόγηση να είναι αρνητική. Οι εργαζόμενοι στην Ευρώπη δεν θέλουμε περισσότερε τέτοιου είδου μεταρρυθμίσει. Δεν θέλουμε λιγότερη κοινωνική ε, κάλυψη. Δεν θέλουμε αυτή τη διακυβέρνηση που όλο και περισσότερο οδηγεί τον φασισμό στο να αναδύεται στην Ευρώπη. Πρέπει η οικονομική σύγκληση και παραγωγική σύγκληση των λαών τη Ευρώπη να είναι η πολιτική μα και να μην είναι η πολιτική μα η αποκένωση τη ε, δημοκρατία και δημοκρατικότητα Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Στη συνέχεια Λάμπερτς. Έχετε τον λόγο. Δυόμιση λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, πρέπει να πω ευθύ εξ αρχή ότι οι πράσινοι αντιλαμβάνονται για να αντιμετωπίσουμε τι προκλήσει του 21ου αιώνα θα πρέπει να συνεργαστούν οι Ευρωπαίοι και να συνεργαστούν και θα πρέπει να έχουμε και ενιαίο νόμισμα. Αυτό συμπεριλαμβάνεται. Πρέπει να διατηρηθεί το ενιαίο νόμισμα. Η ερώτηση είναι ποια μέσα, τα μέσα που διαθέτουμε σήμερα για να εγγυηθούμε τη συνοχή τη Ένωσης, της Οικονομικής και είναι τα δεδειγμένα και τα χρησιμοποιούμε σωστά. Ε, πρώτα απ' όλα, όσον αφορά τη φύση των εργαλείων που διαθέτουμε, είναι σαφές ότι αν έχουμε δημοσιονομική πειθαρχία, ε, ε, και ανταγωνισμό όσον αφορά τα έσοδα, η μόνη μεταβλητή είναι οι δαπάνε. Λοιπόν, να έχουμε δημοσιονομική πειθαρχία όπως ορίζεται σήμερα, χωρίς φορολογική σύγκληση, χωρίς αναρμόνιση φορολογική, θα μας οδηγήσει σε μια μείωση αιώνια του ρόλου του δημοσίου τομέα στην κοινωνία και νομίζουμε ότι αυτό δεν είναι καλό. Θα πρέπει να ολοκληρώσουμε τη δημοσιονομική πειθαρχία με σύγκληση φορολογική. Και εξίσου με τον καθορισμό στόχων περιοριστικών όσον αφορά το περιβάλλον και τα κοινωνικά όταν σαν κυβέρνηση πρέπει να ισορροπήσετε τους προϋπολογισμούς, να συσκελίσετε τον προπολογισμό, να μειώσετε και τη φτώχεια και τι επιπτώσει των περιβάλλων, χρειάζονται προσαρμογέ άλλε από αυτέ βλέπουμε. Χρειαζόμαστε περιοδική, δημοσιονομική πειθαρχία και κοινωνική πειθαρχία. Το εξάμεινο χρησιμοποιείται ευρέω για να προσφυθούν διαθωτικέ ε, αλλαγέ που έχουν στόχο δύο πράγματα. Μείωση του ρόλου του κράτου και να μειωθεί το άμεσο και έμεσο κόστο εργασία και οι εργαζόμενοι ανταγωνίζονται μεταξύ τους και το τρόπος. Λέμε ότι το εξάμεινο θα χρησιμοποιηθεί ανταυτού σαν ένα μέσο συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών, ούτως ώστε να επιτραπεί μια προς τα πάνω ε, δημοκρατική ε, σύγκληση. Αν θέλουμε λοιπόν αυτό το πακέτο οικονομικής διακυβέρνησης Ευρώπης είναι ένα αναγκαίο εργαλείο αλλά ε, δεν χρησιμοποιείται σωστά και δεν ενδείκνυται για την αντιμετώπιση των σημερινών καταστάσεων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Λάμπρεχτς. Ο κύριος Σοφλίν για ένα μισή λεπτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε. Το να αλλάξουμε τους όρους ε, του οικονομικού συντονισμού είναι άλλη ε, μια προσπάθεια απλά για να σώσουμε ένα νόμισμα που δεν λειτουργεί. Και οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που ακούμε τι σημαίνει επισφαλής απασχόληση και περικοπές μισθών δεν θα λειτουργήσει γιατί η Ελλάδα ποτέ δεν μπορεί να γίνει η Γερμανία και η Ιταλία δεν είναι η Ολλανδία. Ο Νέρονας ως γνωστόν έπαιζε, τραγουδούσε ενώ και εγώ ήταν η Ρώμη. Ε, το ότι δεν καίγεται σήμερα η Ρώμη πραγματικά οφείλεται στην στοικότητα των Ιταλών. Αλλά πραγματικά διαλύεται ο κοινωνικός ιστός σε ολόκληρη την Νότια Ευρώπη. Τα ταλέντα των ανθρώπων είναι ο μεγαλύτερος πόρος που υπάρχει και ε, είναι τραγική σπατάλη η ανεργία και ένα νόμισμα το οποίο δεν λειτουργεί καταλήγει στο να μην έχει δουλειά ο κόσμος. Πολλοί εδώ πέρα στην αίθουσα ανήκουν σε διάφορα όργανα τα οποία εξακολουθούν να υποστηρίζουν ένα νόμισμα που δεν λειτουργεί ενώ γνωρίζουν μέσα τους πως λέω την αλήθεια. Πρέπει επιτέλους να πείτε την αλήθεια, να βάλετε επιτέλους τα συμφέροντα των ανθρώπων πιο πάνω από την λανθασμένη ιδεολογία της ολοένα στενότερης ολοκλήρωσης. Όσοι ξέρετε λίγα πράγματα το αντιλαμβάνεστε αυτό. Δεν μιλάτε εδώ και καιρό έχει φτάσει η στιγμή επιτέλους να αποκτήσετε λίγο ανάστημα. Σας ευχαριστώ. Έχετε μια μπλε κάρτα από τον κύριο Λάμπερτς. Ε, την έχετε. Ναι, έχετε τον λόγο. Κύριο Φλίν, θα συμφωνήσω μαζί σας και με πολλούς άλλους που λένε πως ε, δεν είναι βιώσιμη η τωρινή κατάσταση. Ένα κοινό νόμισμα χωρίς, κοινέ, δημοσιο, χωρίς κοινές δημοσιονομικές, ε, οικονομικές και περιβαλλοντικές πολιτικές δεν λειτουργεί. Υπάρχουν δύο απαντήσεις όμως σε αυτό. Είτε πάμε προς τα πίσω στην διάλυση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης και πάμε πίσω στα ε, κράτη-μέλη ή πάμε σε περισσότερη ολοκλήρωση που θέλουμε εμείς. Τι έχετε να μου πείτε. Απάντηση. Την αλήθεια λέτε. Πράγματι ή το ένα ή το άλλο πρέπει να γίνει. Αλλά δεν υπάρχει το επίπεδο κοινωνικής αλληλεγγύης μεταξύ εθνικών κρατών. Εγώ θυμάμαι τη γερμανική επανενοποίηση και οι δυτικογερμανοί γκρινιάζανε. Αλλά επειδή ενώνονταν με άλλους Γερμανούς, το πλήρωσαν το κόστος, δεν είχαν πρόβλημα, αλλά δεν θα πληρώνουν επάπειρον για τους Έλληνες ή άλλους λαούς της Νότιας Ευρώπης. Εάν υπήρχε κοινωνική αλληλεγγύη, αυτή θα ήταν η απάντηση. Αλλά δυστυχώς πρέπει να ε, επιστρέψουμε στα εθνικά κράτη της μεγάλης μας Υπήρου. Σας ευχαριστώ. Μπάρμπαρα Κάπελ για λεπτό. Äh, Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε τον κύριο Επίτροπο Μοσκοβισή στην Επίτροπο Οικονομισματικών Νομισματικών στα όσα αναφέρθηκαν για την ανάλυση εξάπτυχων και δίπτυχων Τον ρώτησα με πόσο σοβαρό τρόπο αντιμετωπίζεται η εφαρμογή και η υλοποίηση αυτών των μέτρων και της, του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης και τι θα γίνει με κυρώσεις και πρόστιμα αν αυτά ε- θα, θα εφαρμόζονται αυτόματα. Είπε ότι τα παίρνει πολύ στα σοβαρά. Είπε όμως ότι μέχρι το Μάρτιο θα άφηνε περίοδο για την Ιταλία, την ε, Γαλλία και το Βέλγιο για τα προβλήματα που υπάρχουν να αναζητηθεί μια λύση σε αυτά τα προβλήματα. Για μένα είναι αυτό αντίφαση στους ίδιους τους όρους, in Και ρωτώ, τι θα γίνει με αυτούς τους πιο περίπλοκους κανόνες της διακυβέρνησης για το Σύμφωνο Σταθερότητας Ανάπτυξης, τα εξαπλά και δίπτυχα που δεν τηρούνται και τι θα γίνει με την μη τήρηση που δεν υφίσταται κυρώσεις μακροπρόθεσμα. Τι θα γίνει λοιπόν και τι θα αλλάξει μέχρι το Μάρτιο του 2015. Ο Υπουργός ε, της Γαλλίας είπε ότι η Γαλλία θα υποβάλει ένα πρότυπο, ένα, μια πρόταση για μεγαλύτερη ανάπτυξη, ιδιωτικοποίηση και τα λοιπά από πλευράς επιχειρήσεων. Όλα αυτά είναι, θα έλεγα, δεν είναι η σωστή προσέγγιση για την ανάπτυξη. Και η Ιταλία σε σχέση με τη μεταρρύθμιση της αγοράς εργασίας ε, έχει οδηγήσει χιλιάδες ε, διαδηλώσεις στους δρόμους. Τι γίνεται σε σχέση με τη διακυβέρνηση των μέτρων αυτών, την οικονομική διακυβέρνηση όταν δεν τηρούνται τα συμπεφωνημένα και δεν επιβάλλονται κυρώσεις και πρόστιμα όταν δεν τηρούνται. Σας ευχαριστούμε πολύ και τώρα θα λάβει τον λόγο για δύο λεπτά στη συνέχεια Θάλμα άλμα Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρόεδρε κυρίες και κύριοι εδώ το Τούπακ και το Σίξπακ που συζητάμε πιστεύω ότι είναι πρόδειλα τα αποτελέσματα τα οποία είναι θετικά. Αν αναλύσουμε την κατάσταση των χωρών της Ευρωζώνης υπήρξαν σημαντικές πρόοδοι όσον αφορά την εξυγίανση καθώς επίσης και σημειώθηκαν πρόοδοι όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις. Η πλειοψηφία των κρατών ξεκίνησαν ήδη να ε, μαθαίνουν και να εφαρμόζουν αυτές τις μεταρρυθμιστικές ε, ε, πρωτοβουλίες. Οι πιο φιλόδοξες χώρες καταδείχθηκε σε σχέση με την εξυγίανση και οι πιο φιλόδοξε όσον αφορά τα προγράμματα μεταρρύθμισης είναι σήμερα οι χώρε που έχουν μεγαλύτερη ανάπτυξη και είναι σήμερα οι χώρε που δημιουργούν μεγαλύτερη απασχόληση. Αλλά δεν επαρκούν όλα αυτά κυρίε και κύριοι. Πρέπει να συνεχίσουμε οπωσδήποτε. Πρέπει να είμαστε πιο στεναροί και αποτελεσματικοί με τι χώρε εκείνες που δεν τηρούν τα συμπεφωνημένα. Διότι οι χώρε αυτέ ε, έχουν επιπτώσει ε, με τη συμπεριφορά του στι υπόλοιπε χώρε τη Ευρωζώνη. Και επιπλέον όπω είπε ο αντιπρόεδρο, είναι είναι αναγκαίο σε όλη αυτή τη διαδικασία να υπάρχει μέγιστη διαφάνεια. Είναι αναγκαίο σε όλη αυτή τη διαδικασία να υπάρχει μεγαλύτερη νομιμότητα δημοκρατική. Διότι σε μια συγκυρία που είναι αναγκαίο να προχωρήσουμε σε αυτή τη δημιουργία της οικονομικής, νομισματικής και στο τέλος πολιτικής ένωσης είναι όταν οι πολίτες στο τέλος τέλος, οι πολίτες της ζώνης ευρώ θα μπορούν να μην αισθάνονται πιο απομακρυσμένοι από τη ζώνη ευρώ. Και δεν έχω καμιά αμφιβολία ότι η έλλειψη, νομισματι... Ε, η έλλειψη δημοκρατικότητας και ε, νομιμοποίησης είναι αυτό το οποίο τους απομακρύνει. Πρέπει να υπάρξει λοιπόν μεγαλύτερη νομιμοποίηση δημοκρατική και για τα εξαπλά μέτρα και για τα διπλά. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε εμείς πολύ και στη συνέχεια η, κυρία, η επόμενη αγορήτρια η κυρία Τόμας δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όταν ξέσπασε το 2009 η κρίση επίτροπε, είδαμε ότι χρειάζεται νομισματική πολιτική. Απεκαλύφθη η, η πολιτική που δεν λειτουργήσε. Λοιπόν, εισαγάγαμε την τροή κάτω από το Ξάμινο. Αλλά πίσω από αυτές τις λέξεις μια πολιτική. Λιτότητα για τους περισσότερους ε, και τα χρηματοδότηση των τραπεζών. Έξι χρόνια μετά την κρίση βλέπουμε ποια είναι η πραγματικότητα κατά πρόσωπο. Αποτυχία. Οι μακροοικονομικές επιλογές της Ένωσης ήταν εργαλεία λιτότητας, που ήταν καταστροφική λιτότητα. Και εκεί που εφαρμόστηκαν οι κανόνες καταστροφικοί. Η Ευρωζώνη αντιμετωπίζει κρίση ακόμα. Έχει 7 εκατομμύρια παραπάνω ενέργους στην Ευρώπη, ένα τρίτο παραπάνω από όταν ξεκίνησε η κρίση. Το χρέος των κρατών δεν μειώθηκε, το έλλειμμα των επενδύσεων είναι 300 δις ευρώ το χρόνο ε, και έχουμε πληθωρισμό υπάρχει και διαφορά, αύξηση διαφοράς μεταξύ των κρατών μελών. Οι κανόνες σύγκληση οδηγούν στην απόκληση τελικά. Η κατάσταση είναι ε, με πολύ χαμηλά επιτόκια, ε, μεγάλη ρευστότητα διαθέσιμη και έλλειμμα ιδιωτικών επενδύσεων που καθυστερεί την ανάπτυξη. Και θέλετε να μείνει αυτή η διακυβέρνηση που εμποδίζει τα κράτα οι μέρη να ανακάμψουν. Και δεν λύνεται το πρόβλημα των χωρών που έχουν κρίση. Λοιπόν, στο σχέδιο το επενδυτικό χρειάζεται μια ευελιξία όσον αφορά το δημόσιο έλλειμμα. Χρειάζεται πλέον να αλλάξουν τα ευρωπαϊκά εργαλεία διακυβέρνησης, να προωθηθούν οι επενδύσεις, να υπάρχουν κοινωνικά κριτήρια, κυρίως το θέμα της απασχόλησης, να υπάρξει φορολογική σύγκληση. Χρειάζονται μακροοικονομικοί κανόνες σίγουρα και οι κανόνες θεσπίζονται για να γίνονται σεβαστοί, υπό τον όρο να αποδίδουν τα μέτρα. Και οι κανόνες σύγκλησης του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης μέχρι τώρα οδήγησαν στην ύφεση, στο χάος και στην διαφοροποίηση των κρατών. Σας ευχαριστούμε πολύ και στη συνέχεια Φων Στόρχ, παρακαλώ. Κυρία Φων Στόρχ, παρακαλώ. Ναι, Ευχαριστώ και ιδιαίτερα εσάς κύριε Επίτροπε Ντομπρόφσκης. Με εντυπωσιάσατε σήμερα πρέπει να πω δώσατε τον απολογισμό σας για όλα αυτά τα πακέτα μέτρων, το διπλό, το εξαπλό, το δημοσιονομικό και όλα τα, όλες τις δέσμες μέτρων. Απαριθμίσατε τις επιτυχίες λέει που έφεραν όλα αυτά τα μέτρα και όλες αυτές τις επιτυχίες τις σημείωσα εδώ όπως τις απαριθμίσατε σε αυτό το λευκό φύλλο χαρτί. Είναι απόλυτα κενό αυτό το λευκό φύλλο χαρτί, καμία επιτυχία. Βλέπουμε τις επιτυχίες λοιπόν τετραετών μέτρων χαρακτηρίζονται επιτυχίες χωρίς να υπάρχει ένα αριθμητικό στοιχείο που να αναφέρεται. Ούτε ένα αριθμό δεν μας αναφέρεται. Δεν βρίσκεστε εδώ μόνο μπροστά ε, στους ευρωβουλευτές αλλά μπροστά στους 500 εκατομμύρια πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και λέτε ότι αυτές είναι επιτυχίες σας. Είναι πραγματικά χρεοκοπία αυτό. Είναι πραγματικά παινία και η πλειοψηφία αυτού του σώματος ζητεί και εκλυπαρεί τον σεβασμό των κανόνων. Οι κανόνες πρέπει να τηρούν οι κανόνες πρέπει να τηρούνται. Και οι συνάδελφοι ζητούν εδώ τον, την κατάργηση του φορολογικού ανταγωνισμού, ιδιαίτερα φιλελεύθερο μέτρο. Όλα τα μέτρα που αναλαμβάνονται αποτυγχάνουν. Και όταν έχετε την ευκαιρία να μας πείτε ποιες είναι οι επιτυχίες, μας δίνετε ένα λευκό φύλλο χαρτί. Και ενώ φύλλο χαρτί είναι η λαθασμένη πορεία αυτή λοιπόν. Σας ευχαριστούμε. Ο Φιλίπ Ντεμπάκερ, επόμενος. Ε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αυτό το οποίο δεν ακούω εγώ στην συζήτηση είναι το ότι μας αφορά εμάς. Μιλάμε για τα κράτη-μέλη που δεν κάνουν τη δουλειά τους, για την Κομισιόν, για περισσότερη ευελιξία, αλλά θα έπρεπε να είναι κάτι το αυτονόητο να είναι ίσως και λυσμένοι οι προπολογισμοί. Θα έπρεπε τα κράτη-μέλη από μόνα τους να προσπαθούν να εξυγχρονίσουν την ε, οικονομία τους. Αυτό είναι για τις επόμενες γενιές ε, και για τις τωρινές απαραίτητο. Αλλά συζητάμε μόνο για το διπλό και το εξαπλό πακέτο. Πρέπει πράγματι να ενισχύσουμε το διπλό και το εξαπλό πακέτο και την ε, δημοκρατική τους νομοποίηση. Αλλά ένα, από ένα πράγμα δεν μπορούμε να ξεφύγουμε. Πρέπει οι προϋπολογισμοί να είναι ισοσκελισμένοι και η οικονομία μας να γίνει πιο ανταγωνιστική από ό,τι είναι σήμερα. Οτιδήποτε άλλο πραγματικά είναι κίνδυνος για τις επόμενες γενιές. Και πρέπει η Κομισιόν να φροντίσει να δει πώς θα ενισχυθεί το διπλό και το εξαπλό πακέτο για να προχωρήσουμε ξανά στον δρόμο της ανάπτυξης και των θέσεων εργασίας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. ευχαριστώ. ένα λεπτό. Υπάρχει εδώ αυτό το οποίο λέγεται Tupac το να πατήσει κανείς μια σκανδάλη για να σκοτώσει ένα μαύρο είναι λέει ε, ηρωική πράξη. Ε, πρώτα που έχουμε τα ναρκωτικά που διακινούνται και μετά σκοτώνονται, ε, δολοφονούμε τους μαύρους. Φαίνεται ότι εδώ σε σχέση με το ατακράτη του Νότου έχουμε μια ανάλογη κατάσταση. Το σύμφωνο σταθερότητας, το σύμφωνο ανάπτυξης είναι λανθασμένο και δεν μπορεί να δημιουργήσει καμία αλλαγή. Επίσης έχει γίνει η παγκόσμια προσέγγιση που υιοθετεί η Ευρώπη και αυτό είναι ε, αποτυχία. Επίσης, ε, για άλλη μια φορά λέμε στους ε, πολίτες ότι πρέπει να υπάρξει αφέμαξή τους. Το αίμα είναι εκείνο το οποίο θα καθαρίσει την κατάσταση. Και τώρα παρουσιάζονται αυτά σαν ε, ένα πρόσχημα για να νομιμοποιηθεί κάτι το οποίο είναι παράνομο σε σχέση με την κρίση. Γι' αυτό και για να ολοκληρώσουμε σας ε, προσκαλώ να εξετάσουμε σε σχέση με το τι έγινε με τους ε, εξαφανιστέντες και αγνοούμενους. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ και παρακαλώ να μην ενοχλείστε για όταν γίνεται μια τέτοια παρέμβαση και στη συνέχεια έχετε εσείς τον λόγο παρακαλώ. Ευχαριστώ. Δεν νομίζω ότι η απλή αναθεώρηση της οικονομικής διακυβέρνησης αρκεί για να λυθεί η βαθιά κρίση στην οποία ε, ε, βρίσκεται η υπηρεσία μας. Και η ύφεση των τελευταίων ετών δείχνει ότι ε, οι κανονισμοί ευρωπαϊκοί στραγγάλισαν κάθε δυνατότητα ανάπτυξης. Το six pack και το twin pack Ολοκληρώνουμε τραγικό τρόπο με διαδρομή που ξεκίνησε το 1997 με την εφαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Ένα όνομα που σήμερα μοιάζει σαν αστείο, διότι σταθερότητα έγινε μια πολύ επικίνδυνη ισορροπία προς τα κάτω και ανάπτυξη δεν είδαμε καν ίχνος. Καλό τους πολίτες κατά τις διακοπές των Χριστουγέννων να διαβάσουν ίσως κάτι που είπε ένας πρώην υπουργό, ο Τζιζέπε Πεγκαρίνο, μια μελέτη. Ε, που, ε, λοιπόν, που μίλησε με συγκεκριμένα επιχειρήματα παρατέθοντας συγκεκριμένα στοιχεία και προσπαθούμε να δούμε πώς όλοι αυτοί οι κανονισμοί που διαδέχτηκαν ως τον άλλον ήταν αντίθετοι από τους στόχους ε, που βγαίνουν από τις συνθήκες, δηλαδή ανάπτυξη που και απασχόληση. Λοιπόν, θα πρέπει να ξαναφύγουμε από το πνεύμα των συνθήκων ε, και τελικά να ξεφύγουμε από αυτού του κανονισμού οι οποίοι θα την ανάπτυξη, να ακολουθούν το πνεύμα των συνθήκων. Σα ευχαριστώ. Ο Συνοδεινό Γιάννη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εδώ και πέντε χρόνια η κρίση δημοσίου χρέου μαστίζει χώρε τη Ευρώπη και ιδιαίτερα του Νότου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αφενό απέτυχε να αντιμετωπίσει την κρίση σε πρώιμο στάδιο, αφετέρου απέδειξε με τη στάση τη ότι εντό του ενωτικού πλαισιού ισχύουν δύο μέτρα και δύο σταθμά έτσι υπάρχουν χώρες που κατηγορούν άλλες χώρες για ανευθυνότητα χώρες που επιτηρούν άλλες και που απαιτούν από αυτές ιδρά δημοσιονομική πειθαρχία καταλύοντας κάθε έννοια εθνικής κυριαρχίας και δημοκρατίας. όλα τα μέτρα οικονομικής διακυβέρνησης ιδιαίτερα οι δίπτυχοι και εξάπτυχοι δέσμοι μέτρων αποσκοπούν σε μια ενισχυμένη διαδικασία επιτήρησης σε μια ένα οικονομική φυλακή όπου τα πάντα εξαρτώνται από τους αριθμού και τις στατιστικές εις βάρος των πολιτών των χωρών. σας διαβεβαιώ ότι είναι απολύτω ανόητο να προσπαθήσουμε να πείσουμε του λαού μα ότι όλα γίνονται για το καλό του. δεν μπορεί ο ελληνικό λαό όπω και οι λαοί τη ιταλία τη ισπανία τη πορτογαλία και συντόμω και άλλοι να βυθίζονται σε οικονομική εξαθλίωση επειδή εσεί υποτάσσεστε στι απαιτήσει των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και των τραπεζικών συμφερόντων. επιτέλου α γίνουν πράξη αυτά που υποσχόμαστε βιώσιμη ανάπτυξη κοινωνική ευημερία καταπολέμηση ανεργία ω ευρώπη των λαών και όχι των οικονομικών μεγεθών. ευχαριστώ δύο λεπτά You have the floor. τον λόγο κύριε Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, θα ήθελα καταρχάς να πω ότι το σύστημα δημοσιονομικής πειθαρχίας κατά την άποψή μου είναι ένα στοιχείο απαραίτητο στα πλαίσια της νομισματικής ένωσης. Τα κράτη-μέλη διατηρούν την αρμοδιότητα αλλά δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο φορολογικό. Χρειάζεται ένα σαφές σύστημα. Να επενθυμίσω ότι η κρίση στην Ευρώπη ξέσπασε όχι διότι εισαγάγαμε το ευρώ αλλά διότι σε κάποια κράτη-μέλη ε, υπήρχαν υπερβολικά χρέη δεν υπήρχε ε, κανένα καθήκον δεν προβλεπόταν από νομοθετικό κείμενο να χρεωθούν. Πρέπει να πω ότι η εμπειρία από τη λειτουργία του Twin Pack και του Six Pack δείχνει ότι χρειάζεται να γίνει προσαρμογή. Είναι περιπλοκότατα, δυσκολότατα συστήματα, όχι για τους εμπειρογνώμονες αλλά για την κοινή γνώμη. Και αυτού του είδους τα συστήματα ε, μπορούν να ερμηνευθούν ποικιλόμορφα Παραδείγματο χάρη, ακούμε ατέρμονες συζητήσει όσον αφορά το βαθμό προσαρμογής των συστημάτων. Θα πρέπει να πλουστευτούν τα συστήματα ώστε να είναι πιο ευληπτά και για τον απλό πολίτη να είναι κατανοητά. Δεύτερο να πω ότι το σύστημα είναι πολύ πολιτικό, έχει μια πολιτική πτυχή υπερβολική. Δηλαδή αφορά όχι μόνο την πολιτική διαδικασία του ελλείμματος, του υπερβολικού ελλείμματος, αλλά αφορά εξίσου τις θεσμίες για την κατάθεση ορισμένων εγγράφων. Πιστεύω ότι αν υπάρχουν νομικοί κανόνες δεν θα πρέπει πλέον να αποτελούν αντικείμενο πολιτικής συζητήσεως αυτοί οι κανόνες. Εν συνεχεία, έχουμε αυτό που αποκαλούμε ιδιοκτησία, ownership. Είναι απαράδεκτο η πολιτική ε, άνδρες να δα, δακτυλοδεικτούν τις Βρυξέλλες. Ότι οι Βρυξέλλες επιβάλλουν τη δημοσιονομική πειθαρχία. Όχι, η δημοσιονομική πειθαρχία θα πρέπει να θεσπίζεται από την εθνική νομοθεσία με συνεκτικό τρόπο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έτσι οι πολιτικοί θα είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόζουν και την εθνική νομοθεσία. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Ροζάτη. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα παρατηρήσατε πως έχουμε ένα μικρό προβληματάκι με τους ε, πίνακες και το τι δείχνουν. Ε, η κυρία Τόια έχει τον λόγο. Κυρία Τόια. Σας βλέπω, σας βλέπω. Ναι, ναι. Οι... Ίσως μπορούν να μας βοηθήσουν οι υπηρεσίες των κοινοβουλευτικών ομάδων. Θα ανακοινώνω πάντα και τους δύο επόμενους. Λοιπόν, μετά την κυρία Τόια θα μιλήσει ο κύριος Φαντάλεν και μετά ο κ. Στόρβαλτς. Κυρία Τόγια, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, αν οι διατάξει του Twin Pack και του Six Pack θεσπίστηκαν για να συγκρατηθεί το χρέο και να ευνοηθεί η ανάπτυξη και αν η σημερινή κατάσταση είναι τόσο αρνητική από όλε τι απόψει, σα ερωτώ, τι πρέπει ακόμα να συμβεί για να καταλάβετε ότι κάτι δεν πάει καλά. Εμείς δεν θέλουμε να παραβούμε τους κανόνες, το λέω σε όλους τους ανήσυχους συναδέλφους. Θέλουμε να είναι χρήσιμοι και λειτουργικοί κανόνες και να πετυχαίνουν το στόχο. Θέλουμε μια ευελιξία ευφυή, δηλαδή χρήσιμη, με καλές επενδύσεις, με σωστές δαπάνες, ούτως ώστε να μπορεί να αναπτυχθεί το ΕΠ. Ευελιξία δεν το αντίθετο της αξιοπιστίας, όπως κάποιοι είπαν αυτές τις μέρες είναι αντίθετο από την ακαμψία, την αντιπαραγωγική που μας οδήγησε μέχρι τώρα. Η εφαρμογή θα πρέπει να είναι λογική, ευέλικτη ε, και θα πρέπει εάν θέλουμε λογιστικά να κυβερνούμε, θα ας μας ε, κυβερνά ένας υπολογιστής και όχι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 40% των Ιταλών που ψήφισαν στις τελευταίες ευρωεκλογές στην Ιταλία ζητούν ευελιξία όχι μόνο για το σχέδιο Juncker αλλά για τη συγχρηματοδότηση των προγραμμάτων που εγκρίνονται την Ευρωπαϊκή Ένωση εντός του προγράμματος για το 2020. Αρκούν αυτές οι μανιακές ιδεολογίες που καλύπτουν τις φορολογικές πολιτικές, τις πολιτικές για την ανάπτυξη και τι επιθέσει κατά τη Ιταλία. Κάποιοι λένε τι κάνει η Ιταλία. Να σα πω τι κάνει η Ιταλία. Η Ιταλία κάνει τι μεταρρυθμίσει η Ιταλία σέβεται τους κανόνες. Θέλει όμως μια πολιτική συνετή, ευφυή, πολιτική, οικονομική που βοηθά να πετύχουμε το στόχο. Δεν θέλουμε να ευνοηθούμε. Θέλουμε ευφυή, πολιτική, αυστηρή ε, που να είναι και μακρόπνοη. Ευχαριστούμε κύριε Τόγια. Ο κύριος Φαντάλεν για 1,5 λεπτό. Μετά Τόρβαλτς και Κατρούγκαλος. Κύριε Φαντάλεν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, η αναθεώρηση του διπλού και του εξαπλού πακέτου έρχεται σε μια πολιτικά ευαίσθητη στιγμή. Θέλουν οι ελίτ να μας κάνουν να πιστέψουμε πως ε, έχει περάσει η ευρωπαϊκή κρίση. Αλλά έχουμε εδώ πέρα δύο βασικά προβλήματα. Πρώτον, η Γαλλία, η Ιταλία και το Βέλγιο δεν έχουν τα οικονομικά τους σε τάξη τα δημόσια οικονομικά τους και ε, για πολιτικούς λόγους εξαιρούνται από τα κριτήρια. Βλέπετε λοιπόν εδώ πέρα πως ε, υποβαθμίζεται η αξιοπιστία της ε, διακυβέρνησης της Ευρωζώνης. Δεύτερον υπάρχουν χώρες στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση οι οποίες τελικά δεν ταιριάζουν εδώ πέρα. Βλέπετε πως οι κύριοι Σαμαράς και Βενιζέλος προκήρυξαν ε, πρόορες εκλογές και από ό,τι φαίνεται η Ελλάδα θα είναι σε καλύτερη κατάσταση εκτός του ευρώ θα μπορούν να υποτιμήσουν και θα έχουν πραγματικά ελπίδα για το μέλλον. Γιατί από ό,τι φαίνεται το βάρος που σηκώνει η χώρα μέσα στην Ευρωζώνη είναι μεγαλύτερο από αυτό που έπρεπε να σηκώσει ο Άτλαντας στις πλάτες του. Έχουμε πάρα πολύ ψηλή ανεργία και κάποιες ευρωπαϊκές οικονομίες θα πάνε πάρα πολύ καλύτερα εκτός της Ευρωζώνης από ό,τι τα πηγαίνουν τώρα. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Φαντάλεν. Ελπίζω να μην γίνουν λάθη. Λοιπόν, το Τόρβαλτς τώρα, μετά ο κύριος Κατρούγκαλος και μετά... Λοιπόν... Τόρβαλς για ένα λεπτό παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ο στόχος αυτού του εγχειρήματο με τα εξάπτυχα και δίπτυχα ήταν η σταθεροποίηση των οικονομικών συστημάτων. Τα αίτια ήταν σαφή. Προφανώς ε, οι χώρες της Ευρώπης σχεδόν συστηματικά παραβίαζαν τα όσα ίσιαν και ζούσαν πάνω από τις δυνατότητες τους ε, και έζησαν έτσι τα καλύτερα χρόνια με υπερχρέωση αλλά οδηγήθηκαν σε ένα αρνητικό τέλος όλα αυτά. Ελπίζουμε ότι θα επανέλθουν οι καλές ε, οικονομικές συγκυρίες. Όμως αυτό δεν έγινε. Δημιουργήθηκαν χρέη. Χρέη τα οποία είναι αφόρητα και δεν μπορεί κανείς να συνεχίσει έτσι υπήρξε και τεχνολογική εξέλιξη, παγκοσμιοποίηση ταυτόχρονα και ιστορικά βλέπουμε ότι οδήγησαν όλα αυτά οι τράπεζες και ο κόσμος των χρηματοοικονομικών να αποκτήσουν υπερβολική εξουσία και το κεφάλαιο όπως ε, συνέβη αυτό και με τα όσα είχαν γραφεί ήδη το 1910 ε, ε, άσκησε αυτό τον αρνητικό ρόλο. Πρέπει να σκεφτούμε τι θα κάνουμε τώρα για να μπορέσουμε να εξέλθουμε από αυτή την κρίση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Τόρβατς. Ακολουθεί ο κύριος Κατρούγκαλος. Ένα λεπτό. Μετά ο συνάδελφος Μάκ και μετά Γκόλνης. Ο κύριος Κατρούγκαλος τώρα παρακαλώ. Επίτροπε, ομολόγησε κάποιες αδυναμίες ε, του πακέτου αυτού η, η Επίτροπη, όπως περιορισμένη διαφάνεια. Θα μπορούσε επίσης να πει ότι άτυπες ομάδες χωρίς λογοδοσία όπως το, ε, ε, η Ευρωομάδα, Eurogroup, έχουν αναλάβει υπερβολικές εξουσίες. Καθώς επίσης ε, και πολλούς άλλους λόγους. Όλες αυτές οι πτυχές είναι σημαντικές καθώς δείχνουν ότι υπονομεύεται η νομισματική και οικονομική κυριαρχία των κρατών μελών χωρίς να υπάρχει υποκατάσταση με άλλα μέτρα. Αυτό βλέπουμε σε σχέση με το ευρώ αντί να αναγνωρίσουμε ότι η λιτότητα είναι αντιπαραγωγική, επιβλήθηκαν περισσότεροι περιορισμοί και περικοπές που θα οξύνουν τη στασιμότητα και θα αυξήσουν την ανεργία και θα υπάρξει ο διαχωρισμός των κρατών μελών σε χώρες ε, που θα έχουν υπερβολική υπερχρέωση και άλλες που θα είναι χώρες χορηγή. Πρέπει να υπάρξει η ενεργοποίηση του ευρωπαϊκού κοινωνικού προτύπου. Και όταν θα γίνουν εκλογές οι Έλληνες είναι εκείνοι που θα ανατρέψουν την κατάσταση πρώτη. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε συνάδελφε Κατρούγκαλε και στη συνέχεια ο κύριος Μακ. Ένα λεπτό. Μετά ο συνάδελφος Γκόλνης. Ο κύριος Μαχ παρακαλώ τώρα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ πρόεδρε, συνάδελφε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι τώρα έχουμε καλύτερους κανόνες. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι κανείς δεν συμμορφώνεται με αυτούς τους κανόνες. Πάρτε τη Γαλλία επί παραδείγματι. Πάνω από 4% του ΑΕΠ είναι το έλλειμμά της και όλοι ε, υποκρίνονται σαν να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και αν κάποιο προσπαθεί να εφαρμόσει τους κανόνες σας, είναι ει βάρο ε, της ανάπτυξης και δημιουργείται και υψηλή ανεργία. Μια λανθασμένη πολιτική απόφαση ήταν η εισαγωγή του ευρώ και αυτή οδήγησε σε άλλη εσφαλμένη πολιτική απόφαση, δηλαδή την επιβολή αυστηρών ε, κανόνων οικονομικών δεν λειτουργούν όλα αυτά. Και απευθύνω έκκληση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παρακαλώ, τροποποιήστε τη συνθήκη ούτω ώστε να μπορεί κανείς να βγαίνει από το ευρώ. Ξέρετε ότι στην Ελλάδα και στην Ιταλία υπάρχουν πολιτικά κόμματα που δεν θέλουν το ευρώ. Λοιπόν πρέπει να τους δώσουμε τη δυνατότητα να το κάνουν αυτό. Και η τσεχική δημοκρατία δεν χρειάζεται να μπει στην ευρωζώνη. Ευχαριστούμε κύριε Μαχ. Μία ερώτηση δέχεστε κυρία Μπέρες. Παρακαλώ έχετε τον λόγο κυρία Μπέρες. Ε, Αγαπητέ συνάδελφε, δεν αναγνωρίζετε τη δυσκολία του ότι κάποιοι κανόνες έχουν συντονιστεί κυκλικά οι κανόνες με την οικονομία και δημιουργεί προβλήματα στις χώρες να προσαρμοστούν και είναι προς όφελος όλων και εκείνων που έχουν πλεόνασμα και ε, ο κ. Δράγκη μας ζητά να κινητοποιήσουμε τη γενική ζήτηση στην Ευρωζώνη. Τι έχετε να πείτε πάνω σε αυτό. Κύριε Μάχα, έχετε τον λόγο. Σας ευχαριστώ. Αν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πει ότι θέλει να δώσει κίνητρα για την οικονομία. Αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει ότι σε σχέση με το μονοπόλιο που έχει για την νομισματική πολιτική θα κάνει κατάχρηση της κατάστασης και θα υπάρξει πληθωρισμός και αυτό εις βάρος όλων των άλλων. Εκτός αν θα έπρεπε να επιτρέψουμε στις ε, χώρες αυτές να επιτρέψουμε να εγκαταλείψουν την Ευρωζώνη γιατί δεν μπορούν να ταιριάξουν σε αυτήν. Ευχαριστούμε συνάδελφε Μαχ αγαπητοί συνάδελφοι, ζητώ συγγνώμη που σας επιβαρύνω, αλλά έχουμε τώρα χειροκίνητο τον κατάλογο και καλό θα ήταν από πλευράς των κοινοβουλευτικών ομάδων να αναφερθεί ότι δεν αληθεύει ο πίνακας στι οθόνε. Υπάρχει εδώ, υπάρχει κάποια έλλειψη λοιπόν. Για 1,5 λεπτό ο συνάδελφος Γκόλνης μετά Σολοσάννα και μετά Ο κύριος Γκόλνης παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε Πεντομπρόφσκης, Θεωρούσα θα είναι δίπλα σας ο κύριος Μοσκοβίτσι ο Επίτροπος. Δεν μπορούμε ότι όταν ήταν ε, Υπουργό Οικονομία στην Γαλλία ότι συνέβαλε πολύ για να απορροφηθεί το έλλειμμα, αλλά με λένε ότι ε, τα, τα γαλματίδια στο Μουσείο του Παρθενώνα στην Αθήνα. Ε, λοιπόν, θα μπορεί να δει και εδώ τους πίνακες όταν έρθει και τις εικόνες του Χριστού κλπ. Ας έρθουμε λοιπόν στα πιο απλά θέματα. Το Six Pack και το Twin Pack είναι ένα σύστημα περιοριστικών μέτρων που θέτουν δημοσιονομική πολιτική των κρατών μελών υπό τον έλεγχο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πολλοί ομιλητές υπογράμμισαν τον περίπλοκο χαρακτήρα και την αποτυχία του συστήματος που χρειάζεται μεταρρύθμιση να καταργηθεί ακόμα καλύτερα. Α, αν παραμείνει ε, οι διατάξεις που επικύρωσαν κακό στα κράτη-μέλη όπως το, τη συνθήκη για τη σταθερότητα, για το συντονισμό και τη διακυβέρνηση όλα αυτά θα συνεχίσουν τα προβλήματα. Ακούσαμε τον κύριο Γιούνκερ που διακήρυσε ότι όλα αυτά μπορούν να εφαρμοστούν ευέλικτα προσπαθώντας να καθησυχάσει τις διαμαρτυρίες του Κοινοβουλίου και ακόμα περισσότερα τις διαμαρτυρίες των ευρωπαϊκών λαών, διότι τα αποτελέσματα είναι γνωστά. Είναι η καταστροφή ε, όλων των συστημάτων του κοινωνικού ιστού και του παραγωγικού μηχανισμού. Άκουσα τον συνάδελφο Λαμπέρτες που έλεγε ότι θα πρέπει να γίνει προς τα άνω ο συντονισμός. Δεν χρησιμεύει αν γίνει προς τα πάνω στην Ευρώπη, αν είναι χτίς σε όλους τους ε, του ανταγωνισμού του αχαλήνου του. Ε, σας ευχαριστούμε συνάδελφε ο συνάδελφος Ιάν, μετά Φερνάντες. Ο κύριος Ιάν. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Έχουμε ένα σύστημα οικονομικής διακυβέρνησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση που λειτουργεί. Για την ώρα το πρόβλημα δεν είναι η κατασκευή του συστήματος αλλά αντίθετα το πρόβλημα ε, ε, αφορούν την εφαρμογή του συστήματος διακυβέρνησης. Πρώτα απ' όλα τα εθνικά κοινοβούλια σε κάποια κράτη-μέλη δεν έχουν συμμετάσχει στην όλη διαδικασία ούτως ώστε να καθορίσουν τα αναγκαία εθνικά μεταρρυθμιστικά προγράμματα. Τα προγράμματα της σύγκλησης ή σταθερότητας που ε, διαβιβάζονται από τις, κρατικές, από τις εθνικές κυβερνήσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Λοιπόν, αν κάποια κράτη-μέλη συμφωνούν με τις συστάσεις σχετικά με την αλλαγή των δημοσιονομικών πολιτικών, παρόλη τη συμφωνία τους, τα κράτη-μέλη δεν λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα τόσο ώστε να εφαρμόσουν στην πράξη τις συστάσεις που γίνονται. Τέλος, υπάρχουν δημόσιες ε, διακηρύξεις όσον αφορά την ανεπάρκεια της ευελιξίας στο Six Pack και στο Twin Pack. Από την πλευρά μου θεωρώ ότι δεν είναι το σύστημα οικονομικής διακυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Ενώσεως που δημιουργεί τα προβλήματα, αλλά το πραγματικό πρόβλημα είναι η μείωση ανταγωνιστικότητας κάποιων κρατών μελών και η έλλειψη σταθερότητα όσον αφορά τις πολιτικές που θα εφαρμοζόταν που θα μπορούσαν να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα, την παραγωγικότητα μέσω επενδύσεων, σωστών επενδύσεων και εφαρμογής των τεχνολογικών πρόοδων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Στόλογιαν. Δέχεστε μια ερώτηση από τον ε, κύριο Σάνι. Παρακαλώ. Θα ήθελα να ρωτήσω τον συνάδελφο, πιστεύει πραγματικά ότι η οικονομική διακυβέρνηση Ευρωζώνης λειτουργεί όταν μέχρι το 2013 μόνο τέσσερις χώρες από τις 17 ε, σεβόταν τα κριτήρια του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Πιστεύω ότι αντί να ε, μιλάμε για να ακουγόμαστε θα πρέπει καλύτερα να εξετάζουμε τα αριθμητικά στοιχεία και τα, τις στατιστικές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτησή σας. Όταν είσαι μέσα στο δημόσιο χρέος, έχεις χάσει την ανταγωνιστικότητα σου, έχεις μόνο μια λύση, την αναδιάρθρωση. Και για να γίνει αυτό χρειάζεται αλληλεγγύη. Δηλαδή, οι εταίροι σα να μπορούν να σου διαθέσουν τον αναγκαίο χρόνο να κάνει αναγκαίε μεταρρυθμίσει και να κάνει όλα όσα χρειάζονται στη χώρα τη συγκεκριμένη. Ευχαριστώ, κύριε Στόλογεν. Για 1,5 λεπτό ο κύριος Φερνάντες, μετά ο Σούλικ και μετά ο κύριος Γκουόγκα. Ο κύριος Φερνάντες παρακαλώ έχει τον λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Η οικονομική κρίση του 2010 την άνοιξη κατέστησε σαφή τα προβλήματα τα οικονομικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης που χρειαζόντουσαν μια καλύτερη οικονομική διακυβέρνηση. Είχαμε τα εξάπτυχα και δίπτυχα μέτρα που σήμερα συζητούμε και για τον έλεγχο της οικονομικής διακυβέρνησης των κρατών μελών. Ωστόσο όμως για την οικονομική κρίση του πρώτου εξαμήνου του 2012 όταν άρχισε η εξέλιξη αυτή με σοβαρά προβλήματα έπρεπε να έχουμε μια κοινή οικονομική πολιτική ε, σχέδιο από το οποίο είχαμε την Τραπεζική Ένωση. Βρίσκεται στα σπάργανα αυτό το εγχείρημα. Χρειαζόμαστε μια ε, Ευρωπαϊκή Οικονομική Ένωση ε, σταθερή και γι' αυτό βλέπουμε ότι όλα αυτά τα μέτρα είναι σε εθνικό επίπεδο. Δεν μπορούμε να αναλύσουμε την ε, οικονομική κατάσταση κάθε χώρα, εξετάζοντα μόνο τι επιπτώσει των εθνικών προπολογισμών στα κράτη-μέλη. Πρέπει να εσωτερικοποιήσει η Ευρώπη τα αποτελέσματα αυτή τη ε, ε, οικονομική διακυβέρνηση για την Ευρώπη και όχι μόνο για τα κράτη-μέλη. Πρέπει να αναθεωρηθούν λοιπόν αυτοί οι κανόνε στο σύνολο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, για να έχουμε μια συνολική επικέντρωση των προβλημάτων προβλημάτων σε σχέση με τα προβλήματα των κρατών μελών. Και χρειαζόμαστε την εφαρμογή του Συμφώνου Ανάπτυξη και Σταθερότητα. Όχι μόνο για να υπάρχει καλύτερη αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα, αλλά για να ενταχθεί αυτή η ευρωπαϊκή ανάλυση σε αυτό το συνολικό, σφαιρικό επικέντρο, ε, τρόπο επικέντρωση για τα προβλήματα του συνόλου τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριε Ντομπρόφσκη, δεν μπορούμε να πούμε ότι λειτουργεί αυτό το σύστημα που έχουμε σήμερα. Δεν λειτουργεί σωστά. Χρειαζόμαστε ένα ευρωπαϊκό εγχείρημα οικονομική διακυβέρνηση. Σε Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. ευχαριστούμε κύριε Φερνάνδες. Για 1,5 λεπτό Σούλικ, μετά Γκουόγκα και μετά ο κύριος Ηλικιώτης. Παρακαλώ κύριε, έχετε τον λόγο κύριε Σούλικ. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρίες και κύριοι. Το εξαπλό πακέτο ισχύει από το Δεκέμβριο του 2011, τρία χρόνια γεμάτα. εισήχθη ως ε, στήριγμα στο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης γιατί κανείς δεν το έπαιρνε σοβαρά. Ας δούμε λοιπόν τα αποτελέσματα. Στα τρία αυτά χρόνια που υπάρχει το εξαπλό πακέτο ανέβηκαν τα χρέη της Ιταλίας από 110 σε 135% του ΑΕΠ. Στην Ισπανία από το 70% στο 95%, στη Γαλλία από το 80% στο 95%, οι χώρες αυτές δεν παίρνουν στα σοβαρά το εξαπλό πακέτο. Ας δούμε τη Γαλλία. Το 2010 είπε η Γαλλία ότι το 12 θα τηρήσουμε τον ε, στόχο του 3%. Μετά το 12 είπε θα το τηρήσουμε το 15. Το 14 έγινε 2017 και δεν υπάρχει καμία κύρωση. Και τι λέει ο Γάλλος Υπουργό Οικονομικών, ο κύριος Σαπέν, η Κομισιόν δεν έχει δικαίωμα να απορρίψει τον προπολογισμό μας. Η κυριαρχία αυτή είναι δικαίωμα του Γαλλικού Κοινοβουλίου. Και τώρα ο, θα ελέγξει τον προκάτοχό του, τον κύριο Μοσκοβισή που έγινε επίτροπος. Ε, αυτά είναι αστεία. Ευχαριστώ κύριε Σούλη για ένα λεπτό ο κύριος Γουόγκα και μετά ο κύριος Σιλικιώτης και μετά ο κύριος Φέκμαρκ. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε, κύριε Πρόεδρε. Αυτή τη στιγμή η Επιτροπή ΙΜΚΟ συντάσσει μια έκθεση για την καλύτερη ολοκλήρωση και ένταξη της ενιαίας αγοράς στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Η ενιαία αγορά εγώ θεωρώ πως είναι κλειδί για την ανάπτυξη και είναι κάτι στο οποίο θα πρέπει να εστιάσουμε καθώς τα κράτη-μέλη δεν εφάρμοσαν πολύ καλές οδηγίες και συστάσεις. Αυτή είναι η αποτυχία μας. Επίσης, η ετήσια έκθεση για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ε, δεν υπευλήθη από την Κομισιόν. Πού είναι το Κοινοβούλιο θα ήθελε να προτείνει κάποια αναλυτικά, αναλυτικά εργαλεία. Πρέπει με κάποιο τρόπο να μετράμε τις επιδόσεις μας. η μεθοδολογία για να μετρηθεί η μείωση του διοικητικού βάρους. Υπάρχει υπερβολική γραφειοκρατία. Αλλά ας τη μετρήσουμε τουλάχιστον για να ξέρουμε τι πρέπει να γίνει. Επιπλέον θα ήθελα να τονίσω την ε, σημασία της εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, αλλιώς δεν έχει νόημα να μιλάμε για πυλώνα ε, εσωτερικής αγοράς. Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Σας ευχαριστούμε. Για ένα λεπτό συνάδελφος Σιλικιώτης. Μετά Χεκμαρκ. Έχετε τον λόγο κύριε Σιλικιώτη. Αγαπητοί συνάδελφοι, η αξιολόγηση της Κομισιόν είναι πρόχειρη και πολιτικά κατευθυνόμενη ώστε να δώσει το μήνυμα πλήρους επιτυχίας των οκτώ νομοθετημάτων χωρίς προβλήματα στην Ευρωζώνη, δικαιολογώντας έτσι την λιτότητα και τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές. Αξιολογείται ως επίτευγμα η δυνατότητα των κρατών να δανείζονται από τις διεθνείς αγορές αλλά δεν προβληματίζει η στασιμότητα η οποία έχει εισέλθει η ευρωπαϊκή οικονομία την τελευταία εφταετία. Επίσης, αναφέρεται ως επίτευγμα η μείωση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων αλλά δεν γίνεται καμία αναφορά στο κοινωνικό κόστος που έχει η πολιτική αυτή. θεμελιακοί παράγοντες όπω η ύφεση τα υψηλά ποσοστά ανεργίας ιδιαίτερα ανάμεσα στους νέου η φτωχοποίηση του πληθυσμού και η ένταση του χάσματος μεταξύ κέντρου και περιφέρεια απουσιάζουν από την αξιολόγηση της επιτροπής. η αριστερά δεν αποδέχεται η κομισιόν να καθορίζει τη στρατηγική στην οικονομική πολιτική των κρατών μελών. δεν υπάρχει δημοκρατική νομιμοποίηση γι' αυτό. στόχος μας είναι η αξιοπρεπή διαβίωση του ανθρώπου αυτό σημαίνει δυνατό κοινωνικό κράτος ασφαλείς θέσεις εργασίας και έμπρακτη αλληλεγγύη. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Χεκμαξ στη συνέχεια. Έχετε τον λόγο, παρακαλώ. Μικρόφωνο, παρακαλώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ τον Επίτροπο για μια πολύ καλή εισαγωγή. Νομίζω δύο θέματα είναι εδώ πρέπει να τονιστούν. Πρώτα απ' όλα, η οδός προς την υπονόμευση της κοινωνικής ασφάλισης, αυξημένη ανεργία, απολεσθής ανταγωνιστικότητα, κοινωνική ανησυχία, ανησυχία και αναταραχές με τη δαπάνη χρημάτων που δεν έχουμε, δεν είχαμε στη διάθεσή μας. Αν τώρα τα ελλείμματα σε σχέση με την επίλυση και τα ελλείμματα με την, τα, ως κίνητρα της ανάπτυξης σε σχέση με την κατάσταση που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Αν είχε γίνει κάτι άλλο δεν θα την αντιμετωπίζαμε. Δεν είναι τα, οι εξηγιανθήσεις ε, πολιτικές που δημιουργούν προβλήματα. Τα αίτια των προβλημάτων είναι η πεποίθηση ότι μπορεί να επιλύσει κανείς οικονομικά προβλήματα με αυξημένα ελλείμματα και υπερβολική υπερχρέωση. Αυτό είναι το λάθος, αυτή είναι η καταστροφή και αυτό είδαμε. Δεύτερον, η αναθεώρηση του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης που θα μπορούσε να είναι καλό εγχείρημα να το κάνουμε. Αλλά ακόμα περισσότερο πρέπει να γίνει μια πραγματική αναθεώρηση. Δηλαδή όταν θα αντιμετωπίζει τις χώρες με λύματα και χρέη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που δεν εξηγίαναν αυτή την κατάσταση όπως έπρεπε και ανέβαλαν την επίλυση του προβλήματος. Η αξιοπιστία εξαρτάται από το να είμαστε αποτελεσματικοί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να έχει αξιοπιστία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να είναι αξιόπιστη, το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης πρέπει να είναι αξιόπιστο. Αν υπονομεύσουμε αυτή την αξιοπιστία επιτρέποντας τα μεγάλα κράτη-μέλη να διαφέρουν να υπεκφεύγουν όχι μόνο από τις ευθύνες, από τους κανόνες, αλλά και από τις κυρώσεις. Θα κοστίσει όσον αφορά την αξιοπιστία μας. Δεν θα βοηθήσει να επιληθούν τα προβλήματα, θα γίνουν μεγαλύτερα τα προβλήματα, θα βαθυνθεί, επιβαθυνθεί ακόμα περισσότερο η κρίση. Πρέπει να τηρούνται οι κανόνες. Αυτό είναι αναγκαίο. Ευχαριστώ. σε ευχαριστούμε συνάδελφε Χεκμαρκ. Δέχεστε μια ερώτηση της συναδέλφου Ματίας κύριε Χεκμαρκ. Εσείς σας συνάδελφε, επιτρέπετε στη συνάδελφο Ματίας μια ερώτηση. Εντάξει, παρακαλώ κυρία Ματίας, έχετε τον λόγο για την ερώτηση. Ευχαριστώ πολύ. Συνάδελφε Χοκμάρκα κατανοώ ότι πιστεύετε σε αυτούς τους κανόνες και κανονισμούς και αναφέρεστε στην ανάγκη να μειωθεί το χρέος και το έλλειμμα. Όμως το χρέος να μειωθεί με περικοπή των δημοσίων δαπανών, με περικοπή του κοινωνικού κράτους. Ερωτώ, ποια μέτρα είναι εκείνα τα οποία θα οδηγήσουν στο να μειωθεί το χρέος. Γιατί δεν σταματά να αυξάνεται το χρέος και αυτό θα συνεχιστεί ως κατάσταση. Με τέτοια μέτρα πώς θα μειωθεί το χρέος χωρίς να υπάρξει διαθροτική αντιμετώπιση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κυρία Ματίας. Τώρα ο συνάδελφο Σέκμακ να απαντήσει. Κυρία Ματίας, πρέπει να σας πω ότι η απειλή στο κράτος ε, ευημερία και κοινωνικής ασφάλισης ε, προέρχεται από τις πολιτικές που εσείς προασπίζεστε. Πιστεύετε ότι μπορείτε να δαπανάτε χρήματα που δεν έχετε. Και αυτό είναι εκείνο το οποίο πραγματικά οδηγεί στην ανάγκη περικοπών και πολιτικών λιτότητας στα κράτη-μέλη. Και αυτό οδήγησε στην έλλειψη επενδύσεων στη βιομηχανία, στις επιχειρήσεις και στην απουσία δημιουργίας θέσεων απασχόλησης. Δείτε την πραγματικότητα, κοιτάξτε γύρω σας. Πού επιτύχαμε και πού αποτύχαμε. Να είμαστε αξιόπιστοι λοιπόν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε συνάδελφε Χεκμαρ. Μία δεύτερη ερώτηση, μπλε κάρτα θα επιτρέψω. Επιτρέπετε να το κάνω αυτό. Να υπάρξουν αυτές οι δύο ερωτήσεις και θα περιοριστώ σε συναδέλφους που δεν παρενέβησαν. Κύριε Χέκμαρκ, επιτρέπετε μια ερώτηση του συναδέλφου Μονό. Παρακαλώ συνάδελφε Μονό. Μονό ουσί. Ένα Στιγμή παρακαλώ. Να το κάνουμε σωστά. Ο συνάδελφος Μονό παρενέβη λοιπόν. Εντάξει. Ερώτηση του κυρίου Γκόλνης τότε. Γιατί ζήτησε τον λόγο ο κύριος Γκόλνης πρώτος. Επιτρέπετε την ερώτηση του κυρίου Γκόλνης. Παρακαλώ κύριε Γκόλνης. Ευχαριστώ. Συγγνώμη, συγγνώμη και πάλι, λέει ο πρόεδρος. Συνάδελφε Μπερές, σαφώς το εξέφρασα. Δύο ερωτήσεις θα επέτρεπα, είπα. Και αν υπάρχουν πάνω από δύο ερωτήσεις, τότε θα επανορθώσουμε με εκείνους που δεν έχουν παρέμβει. Έχουν παρέμβει δύο, τώρα έχουμε μια πρόσθετη ερώτηση. Ο κύριος Γκόλνης ζήτησε τον λόγο πρώτος και εσείς κύριε μόνο ως τρίτος. Ο κύριος Σέκμακ δέχθηκε την επερώτηση και τώρα έχει ο κύριος Γκόλνης τον λόγο για την ερώτηση. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σύντομος. Πιστεύω κύριε Χόκμαρκ ότι στιγματίσατε τα, δημοσιονομικά, τα δημόσια δημοσιονομικά ελλείμματα. Σε κάποιο βαθμό μπορούμε να δεχτούμε την άποψή σα. Δεν πιστεύετε ότι αυτά τα δημόσια δημοσιονομικά χρέη στην πραγματικότητα είναι συνέπεια κάποιου που είναι ακόμα πιο σοβαρό. Το έλλειμμα των εμπορικών ισοζυγίων. Και αυτά τα εμπορικά ισοζύγια, τα ελλείμματα στα εμπορικά ισοζύγια προκαλούνται από το γεγονός ότι η ευρωπαϊκή αγορά είναι ανοιχτή σε όλες τις χώρες που δεν εφαρμόζουν και διακόπτουν. Σας ευχαριστούμε. ευχαριστούμε κύριε Γκόνης. Ο συνάδελφος Εκμαρκ, παρακαλώ, για να απαντήσει. Μικρό. Μικρόφωνο παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, θα έλεγα στον κύριο Γκόνης, κοιτάξτε γύρω σας τον κόσμο τι γίνεται. Βλέπουμε ελεύθερο εμπόριο, βλέπετε ευημερία Όπου υπάρχει προστατευτισμός οποιοδήποτε είδους βλέπετε έλλειψη ευημερίας, απουσία ευημερίας. Πουθενά στον κόσμο δεν κατάφερε κανείς να αναπτύξει οικονομίες και κοινωνίες έναν πολιτισμό χωρίς ανοιχτό χαρακτήρα αυτών. Δείτε τα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη. Αυτά που αντιμετώπισαν την κρίση είναι εκείνα που έχουν ελεύθερο εμπόριο. Δεν θα σας ζητήσω να ενωθείτε με αυτές τις δυνάμεις, διότι γνωρίζω ότι ανήκετε σε άλλη πτέρυγα. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, σας ευχαριστούμε συνάδελφε Χεκμάρκ. Ευχαριστούμε συνάδελφε Χεκμάρκ. Θα προσπαθήσω να είμαι το δυνατόν δικαιότερος. Σε αυτό ανήκει για μια ερώτηση 30 δευτερόλεπτα να διατίθενται και για μια απάντηση πάλι 30 δευτερόλεπτα. Για 1,5 λεπτό ταν. Μετά καλβέτ σαμπόν και μετά διαρρήκα. Παρακαλώ κύριε Τάν, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, θα μιλήσω Ολλανδικά. Βλέπετε τι γίνεται. Βρέχει, πέφτουν οι κεραυνοί, περιμένουμε σε αυτή την περίπτωση να προσγειωθεί το αεροπλάνο με τον αυτόματο πιλότο. Όχι. Το ίδιο συμβαίνει και τώρα. Αποπληθωρισμός, ε, υψηλή ανεργία, χαμηλή εμπιστοσύνη και ανάπτυξη. Και η Κομισιόν μας λέει πως ε, θα γίνουν όλα καλά με, τον, με το διπλό και εξαπλό πακέτο. Όχι, θα πρέπει να προσαρμοστούμε στις συνθήκες στον άσχημο καιρό που επικρατεί. Δεν γίνεται να πηγαίνουμε με τον αυτόματο πιλότο. Και κάτι άλλο. Ε, βλέπετε εδώ πέρα πως είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα το διαρθρωτικό έλλειμμα. Είναι μια ωραία θεωρία, αλλά δεν έχει ε, πραγματική εφαρμογή. Βλέπετε πως ε, το Διεθνές το Ταμείο και η Κομισιόν και ο ο καθένας έχει τις δικές του εκτιμήσεις οι οποίες διαφέρουν κατά πολύ η μία την άλλη. Θα πρέπει λοιπόν να φροντίσετε να κάνετε κάτι επιτέλους για να οδηγηθούμε σε μία ήπια και ομαλή προσγείωση. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, ο αυτόματος πιλότος τώρα λειτουργεί. Οπότε θα λέω μόνο το επόμενο όνομα, Κάλβε Τσαμπόνη για ε, ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Θα συνεχίσω ισπανικά. Θα ήθελα να παρουσιάσω ε, το όλο θέμα όσον αφορά την αξιοπιστία της Ευρώπης και για το ευρωπαϊκό εγχείρημα. Γι' αυτό έχουμε εκλεγεί όλοι μας το, τα εξαπλά και τα διπλά μέτρα θα πρέπει να αποκτήσουν αξιοπιστία. Ε, δεν είναι... Πρέπει να γνωρίζουμε κάποια κενά που υπάρχουν, ότι υπάρχει διακριτική εφαρμογή κατά χώρα των μέτρων αυτών. Αυτό είναι κάτι που υπονομεύει την ευρωπαϊκή αξιοπιστία. Υπάρχει και η έλλειψη εποπτείας. Διότι είναι λάθος να θεωρηθεί ότι έγιναν θεωρητικές μεταρρυθμίσεις στην Ισπανία. Έγιναν κάποιες περικοπές. Εμβαλωματικά μέτρα εφαρμόστηκαν. Επίτροπε, χρειαζόμαστε να συζητήσουμε περισσότερη Ευρώπη που επαιτείται και για την ενεργειακή αγορά. Δεν το έχουμε αυτό. Και θέλουμε και κεφαλουχικές αγορές. Δεν θα δημιουργήσουμε αλληλεγγύη αν δεν θέσουμε το θέμα και των ευρωομολόγων. Σας ευχαριστώ κύριε Καλβέ Σαμπούν. Τον Λε Ιαρίκ ε, τον Συνάλφο δεν τον βλέπω. Αν έρθει μέχρι να μιλήσει ο κύριο Σάντ θα ξαναπάρει τον λόγο. Εν πάση περιπτώσει ο κύριο Νίτερ Μαΐρ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ αγαπητοί συνάδελφοι. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να πω πως είμαι ικανοποιημένος που συζητάμε αυτό το θέμα, τους κανόνες που εγκρίναμε πριν από λίγα χρόνια, που εγώ θεωρώ πως οδηγούν σε καλύτερες οικονομικές πολιτικές που είναι καλές και για τις χώρες και για όλους εμάς. Επίσης οι πολιτικές αυτές μας βοηθούν να σταματήσουμε την κρίση του χρέους και θα ήθελα να υπενθυμίσω εδώ πέρα στους Βρετανούς συναδέλφους πως η κρίση αυτή δεν επηρεάσει μόνο τις χώρες της Ευρωζώνης αλλά και πολλές άλλες χώρες ε, εκτός ευρώ. Ε, εκπλήσεων που ακούω κάποιους να λένε πως οι κανόνες απέτυχαν. Αυτό το οποίο απέτυχε σίγουρα ήταν οι πολιτικές προ της κρίσης πολλών κρατών. Οι πολιτικές ε, που δημιουργούσαν υψηλότερα ελλείμματα, αύξαναν το χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ, αύξαναν τις δαπάνες ε, και ζητούσαν ανοχή για κακή οικονομική πολιτική. Αν είναι κάποιος υπεύθυνο για την τωρινή υψηλή ανεργία, ε, αυτή είναι η υποπτή κατά την άποψή μου. Τι πρέπει να κάνουμε τώρα. Δεν πρέπει να εστιάζουμε στην αλλαγή του πλαισίου γιατί ε, εγώ θεωρώ πως μέχρι τώρα καλά έχει λειτουργήσει. Πρέπει να προσέχουμε να μην κάνουμε βιαστικές αλλαγές που θα υποβαθμίσουν την αξιοπιστία μας. Ε, υπάρχει, μην ξεχνάμε ότι ε, αύξηση των επιτοκίων κατά 1% σημαίνει αύξηση και του ελλείμματος κατά το ίδιο ποσοστό και επίσης θα επηρεαστεί και η διπισονομική ισορροπία που ενδιαφέρει και τους Βρετανούς ε, συναδέλφους θα συζητήσουμε και άλλα πράγματα, πώς θα μπορέσουμε να κάνουμε τις χώρες να σέβονται τις συστάσεις που τους γίνονται, τι θα γίνει με τις διαρθρωτικές ανισορροπίες ή πώς θα δώσουν περισσότερη προσοχή στις χώρες εκτός Ευρωζώνης. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ κύριε Νίντερ Μάιερ για ένα μισή λεπτό ο κύριος Σαντ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το ρυθμίσει ε, των εξαπλών και διπλών μέτρων ε, προσπαθούν να, να εξασφαλίσουν την εφαρμογή των διαφόρων μέτρων. Χρειάζεται συντονισμένη προσέγγιση για την αξιολόγηση οικονομικών και χρηματοπιστικών αποτελεσμάτων. Δεν υπάρχει ενοποιημένη όμως ε, κεντρική λειτουργία όσον αφορά την Ευρωζώνη. Θα πρέπει λοιπόν να δημιουργήσουμε το σωστό πλαίσιο. Ε, υπάρχουν πολιτικοί παράγοντες που ισχύουν στην Ευρώπη και αφορούν ε, πολιτικό κεφάλαιο ε, που έχει χρησιμοποιηθεί για το ευρωπαϊκό εγχείρημα. Υπήρχε πολυμερής δοσοληψία διαφόρων φορέων που, στη σε διάφορες προσπάθειες και δεν υπάρχει σύγκληση των εθνικών συμφερόντων. Λοιπόν, η βαθμολόγηση, το σύστημα βαθμολογήσεως και των πινάκων βαθμολόγησης, όλα αυτά τα συστήματα ε, καλύπτουν την πραγματικότητα. Ίσως καλύπτονται τα συμπτώματα και όχι τα αίτια του ευρωπαϊκού εγχειρήματος, των προβλημάτων του ευρωπαϊκού εγχειρήματο. Χρειάζεται μεγαλύτερη διαφάνεια. Με μεγαλύτερη διαφάνεια η Ευρωζώνη θα μπορούσε να κινηθεί προς μια πολιτική ομοσπονδιακή δομή. Κάτι πολύ δύσκολο. Λοιπόν, τα εξαπλά και διπλά μέτρα αυτά, τα πακέτα, χρησιμοποιούνται σωστά σε όλα τα επίπεδα, στις διάφορες εθνικές οικονομίες, ανταποκρίνονται στις προσπάθειες για ανάπτυξη της Ευρωζώνης ή αντικατοπτρίζονται εθνικά συμφέροντα κρατών μελών. Δεν μπορούμε να δώσουμε σαφή απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει πρόβλημα συστημικό όσον αφορά το σχεδιασμό των μηχανισμών που έχουμε, που αναπτύχθηκαν μέσω δοκιμών και διπλωματικών δοσοληψιών. Ευχαριστούμε. Ο κύριος παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι υπάρχει ένας κίνδυνος να μπερδέψουμε τους μηχανισμούς με την ουσία, δηλαδή να κάνουμε κριτική στο 2-pack, 6-pack, ουσιαστικά να θέλουμε να σπάσουμε το θερμόμετρο για να μην δούμε τον πυρετό που μας προειδοποιεί ενδεχομένως για μια οικονομική ή δημοσιονομική ασθένεια. Πιστεύω ότι πάμε σε γενικές γραμμές καλά υπάρχουν συγκεκριμένε επιτυχίε, η ιρλανδία βγήκε από το μνημόνιο η πορτογαλία βγήκε από το μνημόνιο λετωνία λιθουανία κάνανε καλή δουλειά και πήραν το εισιτήριο εισόδου στο ευρώ η Κύπρο πηγαίνει σε γενικέ γραμμέ καλά από ό,τι πληροφορούμε Δυστυχώ η χώρα μου η ελλάδα προσπαθεί ακόμα δεν τα έχει καταφέρει. θα σα πω όμω ότι τα προβλήματα τη Ελλάδα, εγώ επειδή ήμουν 35 χρόνια δημοσιογράφο και εκδότη, τα παρακολουθούσα και πριν από το ευρώ και πριν από το two pack και το six pack και πριν από τους μηχανισμούς σταθεροποίησης και θα σας πω ότι σε γενικές γραμμές ήταν τα ίδια δηλαδή δίναμε μεγάλες συντάξεις είχαμε ένα υπερβολικά πλουσιοπάροχο κράτος πρόνοιας που δεν μπορούσε να χρηματοδοτηθεί από τον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας και θα πω στους φίλους μας τους βρετανούς αντιευρωπαίους και ευρωσκεπτικιστές οι οποίοι λένε ότι στην ελλάδα έχουμε τεράστια προβλήματα από το ευρώ ότι παλιά δίναμε συντάξεις στην ελλάδα που ήταν 100 και 120% του τελευταίου μισθού ενώ στο ηνωμένο βασίλειο οι συντάξεις επειδή είχα διαβάσει τα σχετικά ήταν της τάξης του 35 έως 40% του τελευταίου μισθού. επομένως τα προβλήματα προϋπήρχαν δεν μπορούμε να τα αποδώσουμε στο ευρώ. αντίθετα το ευρώ μας διευκολύνει στην αναδιά... σε μια μελλοντική αναδιάρθρωση του χρέους Μα διευκολύνει όπω στην περίπτωση τη Ιρλανδία, στο μέλλον στη μείωση του κόστου δανεισμού ενώ με τα μέτρα που παίρνει ο κύριος Ντράγκη το ευρώ γίνεται λιγότερο ισχυρό και διευκολύνει και την εξαγωγική προσπάθεια χωρών όπω η Ελλάδα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Κίρτσο. Κύριε Κίρτσο, επιτρέπετε μια ερώτηση του συναδέλφου Βάλλη. Μάλιστα. Συνάδελφε Βάλλη, παρακαλώ έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Έχω μια ερώτηση απλούστατη. Πιστεύετε ότι το ευρώ είναι βιώσιμο για τη χώρα σας το ευρώ. Α, λοιπόν, είναι βιώσιμο και το επιτόκιο που πληρώνεται η χώρα σας που είναι περίπου 9% τη στιγμή που είναι υπό οικονομική πίεση, όταν η Γερμανία ίσως πληρώνει ένα 0% εναντί των ελληνικών τόκων. Είναι βιώσιμο το ευρώ χωρίς να υπάρχει ενιαίο επιτόκιο. Συνάδελφε Κίρσο. Το επιτόκιο πληρώνει η χώρα μας, αντίστοιχο με το επιτόκιο που πληρώνει η Ιρλανδία, η οποία διαθέτει τα δεκαετή ομόλογα του δικού της δημοσίου κάτω από 1,5%. Και επειδή η Ιρλανδία πάντων, είναι πολύ δυναμική σαν οικονομία, ας πάμε στα επιτόκια της Πορτογαλίας που είναι συγκρίσιμη με την Ελλάδα τα οποία αυτή τη στιγμή αν δεν κάνω λάθος είναι γύρω στο 2,9%. Είναι γεγονός ότι τα επιτόκια στην Ελλάδα έχουν αυξηθεί αυτή τη στιγμή ακριβώς επειδή οι αγορές δεν είναι σίγουρες αν θα προσπαθήσουμε να ολοκληρώσουμε ε, αυτά που κάνουμε. Ευχαριστούμε πολύ συνάδελφε Κίρτσο. Επιτρέπετε επιπλέον ερώτηση του συναδέλφου Λούκε. Παρακαλώ συνάδελφε, έχετε τον λόγο. Κύριε συνάδελφε, κατάλαβα από αυτά που είπατε ότι το ευρώ θα βοηθούσε λέει την Ελλάδα να αναδιαρθρώσει τα χρέη της. Δεν συμβαίνει περισσότερο το ότι η καλή πίστη των πιστωτών είναι εκείνη που οδήγησε στην αναδιάρθρωση του χρέους σε σχέση με τα 100 δισεκατομμύρια χρέους που παρετήθηκαν από αυτό για να μπορούσε να ε, ξεπληρώσει η, η Ελλάδα το χρέος της. Ευχαριστώ. Αυτή τη στιγμή το χρέος της Ελλάδας είναι δημόσιο, δεν είναι πια στον ιδιωτικό τομέα, άρα έχουμε πολιτική και ηθική υποχρέωση να πληρώσουμε θα πληρώσουμε σε βάθος χρόνου φυσικά. υπάρχει μια συζήτηση να πάει η αναδιάρθρωση του χρέους από 30 χρόνια στα 50 χρόνια για να διευκολυνθούμε αλλά υπάρχουν δύο βασικές προϋποθέσεις να υπάρχουν σταθερά πρωτογενή πλεονάσματα και να γίνουν οι αναγκαίες διαρθρωτικές αλλαγές. επομένως νομίζω ότι έτσι θα βγουν κερδισμένες και οι δύο πλευρές η ελλάδα θα εξυγχρονιστεί και οι πιστωτές της θα πληρωθούν. Ε, σε ευχαριστούμε συνάδελφε Κίτσο. Για 1,5 λεπτό ο συνάδελφος Σάνι παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Λοιπόν, αυτή η συζήτηση όταν την παρακολουθεί κανείς σκέφτηκα παρακολουθώντας την ότι εμείς οι ευρωβουλευτές ή εκπρόσωποι ακόμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όταν σε ένα καφενείο π.χ. ακούνε τέτοιες συζητήσεις και αν θα ρωτούσαν γίνεται κατανοητό από τους πολίτες τι σημαίνει ένα δίπτυχο, τι σημαίνουν τα δίπτυχα μέτρα ή τα εξάπτυχα μέτρα. Ε, αυτή η συζήτηση λοιπόν πρέπει να συνεισφέρει να αποσαφινιστούν αυτά. Ευχαριστώ τους συναδέλφους που συνεισφέρουν να γίνουν αυτά πιο κατανοητά, ότι αυτά τα κείμενα δηλαδή για την αντιμετώπιση της ευρωκρίσης διαδραματίζουν σημαντική, ε, σημαντικό ρόλο. Και υπάρχει και ένα πρόσθετο θέμα που άμεσα ως ερώτημα θέλω να απευθύνω προς τον Επίτροπο. Και αυτό είναι τι είναι αυτό το οποίο γίνεται ώστε ο κοινωνικός διάλογος να μπορέσει να προαχθεί και να βελτιωθεί. Και αυτό διότι έχω την υποψία πρέπει να ομολογήσω ότι αυτά τα μέτρα six pack και two pack δημιουργούν ένα πρόβλημα, έχουν ένα πρόβλημα που δεν κατανοείται από την κοινωνία και γι' αυτό δεν μπόρεσε να γίνει κατανοητό αυτό. Τι θα κάνετε λοιπόν ώστε να υπάρξει ένας πραγματικός κοινωνικός διάλογος για αυτά. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε συνάδελφε Σάνη. Στη συνέχεια η κυρία Χούμπνερ παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Αντιπρόεδρε Ντομπρόφσκης, θα ήθελα να τονίσω τρία θέματα. Το πρώτο, Πιστεύω ότι η ίδια η φύση της οικονομικής διακυβέρνησης μας υποχρεώνει να δούμε πέρα από τον ορίζοντα των εξαπλών και ε, των διπλών μέτρων για μια Τραπεζική Ένωση για παράδειγμα, ακόμα και αν δεν είναι στοιχείο οικονομικής διακυβέρνησης, αλλά μπορεί να συνεισφέρει για τη σταθεροποίηση του συστήματος και θα μπορέσει να δώσει ικανότητα, δυναμικό στην Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση να είναι πιο αποτελεσματική. Ταυτοποιώντας λοιπόν δυνατότητες βελτίωσης, πρέπει να έχουμε αυτή την προοπτική ως προοπτική βελτίωσης. Δεύτερη παρατήρηση, κανόνες έναντι διαδικασιών. Έγινε αναφορά σε αυτό το θέμα. Πιστεύω ότι η οικονομική διακυβέρνηση και το πλαίσιο της πραγματικά δημιούργησε πολλούς κανόνες. Όμως η επιτυχία τους εξαρτάται από την επιλογή των σωστών μέτρων και πολιτικών. Βλέποντας την έκβαση της οικονομικής διακυβέρνησης όμως οι πολίτες δεν διαφοροποιούν μεταξύ των επιλογών πολιτικών και των κανόνων του, του συστήματος. Επιλογών εθνικών φυσικά. Και αυτό δημιουργεί υποψίες για την ε, βιωσιμότητα του συστήματος καθώς και για την αξιοπιστία τη δημοκρατική. Σεβόμενοι τους κανόνες πιστεύω ταυτόχρονα Πρέπει να έχουμε καλύτερες επιλογές πολιτικών που θα είναι κομμένες και ραμμένες για τις ανάγκες μας και να αξιολογήσουμε ακριβώς και το θέμα του πώς θα μπορέσουμε να καλύψουμε την νομιμότητα, το πρόβλημα νομιμότητας. Δεύτερο, για την ανάπτυξη. Οποιαδήποτε οικονομική διακυβέρνηση πρέπει να έχει προοπτική ισχυρή ανάπτυξη και διαφορετικέ ε, πολιτικέ είναι και αναθεωρήσεις είναι αναγκαίε εδώ. Και πρέπει να δούμε εδώ το μηχανισμό για την προαγωγή αυτών των ε, μεταρρυθμίσεων. Μέτρα έχουν προταθεί από, ήδη κατά το παρελθόν και που μέχρι πρόσφατα διαγράφηκαν και εξαφανίστηκαν από την οθόνη του ραντάρ μας. Και φαίνεται ότι από το Δεκέμβριο ξανανοίγεται αυτή η προοπτική. Ελπίζω λοιπόν ότι θα έχουμε στεναρή δέσμευση για τον καταλήτη των διαθωτικών αλλαγών και μεταρρυθμίσεων. Και ελπίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προωθήσει προς αυτή την κατεύθυνση με ενεργό ρόλο προπομπού, πρωτοπόρου. Σα ευχαριστώ συνάδελφε Χίμνερ. Για 1,5 λεπτό, μπαγέ παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Όταν θέλουμε να αξιολογήσουμε τα μέτρα που έχουν συνέπειες μακροοικονομικές τόσο μεγάλες, θα πρέπει να σεβαστούμε τον αξιολογισμό και να υπάρχει και σωστή ανάλυση συνεκτική για το Six Pack και το Twin Pack. Τι ίδια έχουμε, ανακοίνωση τεχνικής φύσης Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αναφέρεται στην ανάπτυξη του δημοσίου χρέους και τελεία και παύλα. Τίποτα όσον αφορά την αξιολόγηση τη συνέπεια, όσον αφορά την οικονομική ανάπτυξη, τίποτα όσον αφορά την ανεργία, τίποτα όσον αφορά τα κοινωνικά δικαιώματα και τίποτα όσον αφορά τη φτώχεια. Λοιπόν, καθημερινά οι περισσότεροι Ευρωπαίοι ε, είναι σαφής αξιολόγηση, ε, το Twin Pack και Six Pack είναι η λιτότητα. Είναι αύξηση της φτώχειας, μείωση των κοινωνικών παροχών, παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων όπως η καθολική πρόσβαση στην υγεία. Ε, στην αξιολόγηση υπάρχει μετά η αντίδραση που είναι κοινωνικά σωστή. Λοιπόν, θα πρέπει να γίνει μοχλός κοινωνικής πρόοδου και ε, ελπίδας η Ευρώπη και να δημιουργηθεί ένα νέο κοινωνικό ε, οκταπλό ε, πακέτο και να μπορεί να παρέμβει ο δημόσιο τομέα εκεί που ο ιδιωτικό τομέα δεν μπορεί. Και το δείχνουν και τα στοιχεία τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τη Τράπεζα Επενδύσεων. Λοιπόν, θα πρέπει να υπάρχει έλεγχο των κερδών μεγάλων κεφαλαίων. Λοιπόν, θα πρέπει να καταπολεμηθεί το κοινωνικό περιβαλλοντικό dumping. Η λιτότητα σήμερα είναι προφανής ότι δεν λειτουργήσε. Ε, προβλεπόταν η κοινωνική ύφεση, αλλά τελικά τα αποτελέσματα είναι πολύ αρνητικά. Λοιπόν, δεν υπάρχει αξιοπιστία στον στρατηγική λόγω των αποτελεσμάτων. Λοιπόν, θα πρέπει λοιπόν να αλλάξει η κατεύθυνση γρήγορα και να επενδύσουμε σε προοδευτικές αρχές και σε κοινωνική δικαιοσύνη. Σας ευχαριστούμε συνάδελφε Μπαγιέ. Συνάδελφε Μπαγιέ, επιτρέπετε μια ερώτηση του κύριου Μανού, παρακαλώ. Πείτε, Μανού. Παρακαλώ, συνάδελφε Μανού, έχετε τον λόγο. Ε, Κύριε Μπαγιέ, συνάδελφε, συμφωνώ απόλυτα με τη δήλωσή σας. Αλλά το κόμμα σας στη Γαλλία και ο πρόεδρός σας τι περιμένει για να εφαρμόσει τους περίφημους αυτούς κανόνες. Αγαπητέ συνάδελφε, ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Δυστυχώ, όταν παίρνετε το λόγο, είναι πάντα για να επικρίνετε του Γάλλου σοσιαλιστέ. Εγώ είμαι Βέλγο σοσιαλιστή ε, και εργάζομαι προ όφελο τη Ευρώπη και για να απαντώ σε απαντήσει εθνικού μετόπου όσον αφορά τον αιώνιο εχθρό του, του σοσιαλιστέ, ε, και την επόμενη φορά θα είναι φιλελεύθεροι. Ευχαριστούμε πολύ. Και όποιο μιλάει γαλλικά θεωρείται Γάλλο, ενώ μπορεί να μην είναι. Για δύο λεπτά, κυρία Κόμη, παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητέ Επίτροπε. Πιστεύω ότι η συζήτηση σημερινή είναι η πιο σημαντική που μπορούμε να κάνουμε υπό την ιδιότητα των Ευρωπαίων βουλευτών και σαν Ευρωβουλευτές εξελέγημεν άμεσα από τους πολίτες για να αλλάξουμε την κατάσταση. Δεν είμαστε εδώ για να κάνουμε διαμαρτυρίες χωρίς προτάσεις. Πρέπει να πετύχουμε σαφείς στόχους, διαφορετικά δεν θα εκπληρώσουμε την εντολή που μας ανέθεσαν οι πολίτες. Λοιπόν, και ο Άγιος Πατέρας στις 25 Νοεμβρίου έκανε σαφές το μήνυμά του. Σαφές μήνυμα το οποίο το βρήκε συμφώνου 99,9% των παρισταμένων στην αίθουσα. Περισσότερη Ευρώπη, μια Ευρώπη πιο ε, δίκαιη και να παραμένει ζωντανή πραγματικότητα της δημοκρατίας. Αυτό το μήνυμα ε, ε, το συνόδευσα με δηλώσει όλε οι ομάδε, με μόνο δύο-τρει που ήταν αντίθετοι. Όλοι συμφωνούσαν. Η οικονομική ανάπτυξη πρέπει να ενώνεται με τη σταθερότητα. Σε μια στιγμή κρίση φτάνει πρώτα η ανάπτυξη. Διαφορετικά ε, δεν μπορεί να πετύχει. Χωρί ανάπτυξη δεν θα έχουμε σταθερότητα. Λοιπόν, και αν για ανάπτυξη πρέπει να χρησιμοποιούμε μεγαλύτερο χρέο μόνο, μόνο και λέω μόνο και, και σαν Ιταλίδα καταλαβαίνω το πώς σας μπλέκω με αυτά που λέω. Για επενδύσεις, γιατί δεν γίνονται, εγώ είμαι πεπισμένη ότι οι επενδύσεις είναι το εφαλτήριο της ε, ανάπτυξης. Και αυτό είναι κάτι που δημιουργεί πραγματικά θέσει εργασία. Εγκρίνω πλήρω το πρόγραμμα Juncker για τη Φορολογική Ένωση. Ε, στην Ιταλία θα λυνόταν πολλά προβλήματα βλέποντα τη φορολόγηση που έχουμε. Ε, Εμεί, οι Ιταλοί βρίσκονται, διαμαρτύρονται το σύμφωνο σταθερότητα σε Ιταλία, αλλά πολύ συχνά ε, κοιτάει κανεί αλλού και στο σπίτι του. Θα πρέπει να τακτοποιήσουμε στα σπίτι μα λογαριασμού, τροποποιώντα το σύμφωνο σταθερότητα στο εσωτερικό, που δεν επιτρέπει στου δημάρχου να ξοδεύουν τα χρήματα που έχουν. Συζητείτε και εδώ κλείνω. Η ανεργία στη Γερμανία όπου υπάρχει το ευρώ, η ανεργία στην Βρετανία όπου δεν υπάρχει το ευρώ και σε αυτή την περίπτωση υπάρχουν πολύ πιο χαμηλοί φόροι από τους δικούς μας. Και κλείνω λέγοντας ότι λέμε στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και διακόπτεται η ομιλήτρια. Σας ευχαριστούμε συνάδελφε Κόμη. Ακολουθεί ο συνάδελφος Μαυρίδης. μισή λεπτό παρακαλώ. Εγώ με τη σειρά μου απευθύνομαι τόσο στους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσο και στους συναδέλφους μου. Ξεκινώ με μια διαπίστωση που πρέπει να δεν υπάρχει γκρίζο, είναι άσπρο ή μαύρο το όραμα της κοινή ευρωπαϊκής στέγης προϋποθέτει κοινή σύγκληση στο οικονομικό επίπεδο διαβίωσης των ευρωπαίων και οι ευρωπαίοι είναι από το ένα άκρο μέχρι το άλλο άκρο. κατανοώ όσους επιμένουν ότι τα χρέη ενός κράτους μέλους δεν πρέπει να μεταφέρονται στους ώμους άλλου κράτους μέλους. ωστόσο τονίζω ότι στα οικονομικά τα πράγματα δεν είναι zero sum αλλά είναι και προσθετικά δηλαδή μπορούμε μέσα από συλλογική διαχείριση να συναποφασίζουμε κανόνες αλλά αυτοί οι κανόνες δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι απόλυτα ήδη ίδιοι για όλα τα κράτη μέλη. επίσης τονίζω προς τους συναδέλφους μου ότι δεν προσδοκώ πολλά από εκείνους που θέλουν να διαλύσουν την ευρωπαϊκή ένωση. η απογοήτευσή μου όμως είναι από εκείνους που δηλώνουν ότι συμμεριζόμαστε το ίδιο όραμα για την ευρώπη αφήνουν όμω έξω του Ευρωπαίου πολίτε ή ένα μέρο των ευρωπαίων πολιτών είτε είναι στον νότο είτε είναι στο βορρά. και καταλήγουμε λοιπόν να έχουμε country specific recommendations αλλά δεν έχουμε country specific φάρμακο. και ένα συγκεκριμένο παράδειγμα έχουμε τραπεζική ένωση αλλά δεν έχουμε κοινό ενιαίο ε, σχέδιο εγγύησης των καταθέσεων αυτά λοιπόν και αναμένω στην ευαισθησία όλων για τον ευρωπαϊκό Ευχαριστώ κύριε Μαυρίδη. Για δύο λεπτά ο κύριος Φερνάντες. Ευχαριστώ Πρόεδρε, Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, συνάδελφοι. Ο συντονισμός και ο συγχρονισμός καθώς και η μέγιστη δυνατή διαφάνεια είναι θεμελιώδους αξίες για τη διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά και η πρόληψη είναι αναγκαία. Πρόληψη είναι καλύτερη από τη θεραπεία, όπως λένε και οι παροιμίες. Και για μας τους Πορτογάλους αυτό σημαίνει επίσης ότι δεν θέλουμε την Τρόικα. Το διπλό και το εξαπλό πακέτο χρειάζονται για να αυξηθεί η αξιοπιστία της Ευρώπης, των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων θα μας επιτρέψουν να εντοπίσουμε προβλήματα πριν γίνουν ανεπίλητα τα προβλήματα και θα αποφύγουμε ανισορροπίες και διοθωτικά μέτρα θα οδηγήσουν σε υπεύθυνη συμπεριφορά και συνεπώς αλληλεγγύη, η ισόρευση των ελλημάτων και αύξηση των χρεών με μη βιώσιμο τρόπο σημαίνει ότι θα πληρώσουμε όλο το τίμημα. Κυρίως οι μελλοντικέ γενιές θα πρέπει να πληρώσουν το τίμημα. Χρειαζόμαστε μια ευφυή και ευέλικτη ερμηνεία των εξαπλών ε, και διπλών μέτρων και των σχετικών κανόνων. Αυτό σημαίνει ότι η πρόθεση οικονομικής ανάπτυξης και της απασχόλησης και η πρόθεση της ε, ανταγωνιστικότητας χρειάζονται προτεραιότητα χωρίς να υπονομεύεται βέβαια εξοπιστία των υποχρεώσεων που έχουμε αναλάβει. Πέραν αυτών, η οικονομική και κοινωνική συνοχή και η εδαφική συνοχή ε, είναι πράγματα που μας προβληματίζουν. Και μια ευφυής και ευέλικτη ερμηνεία των εξαπλών και διπλών αυτών μέτρων θα επιτρέψουν να ληφθούν όπως αυτές οι πτυχές. Ευχαριστώ πολύ κύριε Φερνάντες. Ένα μισή λεπτό. Ο κύριος Ντάντη παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε, συνάδελφοι. Είναι προφανές ότι η ευρωπαϊκή οικονομική governance, διακυβέρνηση, λέει στα αγγλικά ο μιλητής, θα πρέπει να αλλάξει πλέον. Η κατάσταση είναι πλέον επικίνδυνη, υπάρχει διαφθρωτική ανεργία, υπάρχουν κάποιοι πολύ εύθραυστοι ρυθμοί ανάπτυξης και το βήμα Juncker είναι ένα βήμα μικρό, ένα βήμα δήλο, το οποίο θα πρέπει ε, ακόμα να συγκεκριμενοποιηθεί αναζητούμε την προτεραιότητα φυσικά της ανάπτυξης. Αυτό σημαίνει βελτίωση της οικονομικής διακυβέρνησης. Είναι μια καλή ευκαιρία, ίσως είναι η τελευταία ευκαιρία για μια Ευρώπη που δύσκολα οικοδομήσαμε και η οποία λόγω των μειοπικών οικονομικών πολιτικών κινδυνεύει να την αχθεί στον αέρα όπως φαίνεται και στα συμπεράσματα του Συμβουλίου τον μήνα Ιούνιο. Η ευελιξία αυτή δεν αρκεί από μόνη της, δεν μπορεί να είναι μια απλή παραχώρηση, πρέπει να είναι μια θεμελιώδη στρατηγική. Τα κράτη-μέλη πρέπει να την επιδιώξουν σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα. Και δεν μπορούμε να βασίσουμε όλες τις δυνατότητες ανάπτυξης στο σχέδιο Juncker, εάν παράλληλα δεν μπορεί να υπάρξει μια πίεση προς πιο ευφυείς μορφές επενδύσεων. Εμείς δεν μιλάμε αφηρημένα εμείς θέλουμε ε, να προσπαθήσουμε να βασιστούμε και στο σχέδιο Juncker αλλά να οδηγηθούμε σε μια πραγματική οικονομία για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Ευχαριστώ κύριε Ντάντη. Για δύο λεπτά η κυρία Παύνοβα. Ευχαριστώ Πρόεδρε Επίτροπε. Θα πρέπει να σας πω ότι ε, σε ό,τι αφορά ε, τα ε, μέτρα αυτά που λαμβάνονται είναι πρωτοφανής η κατάσταση. Ε, όταν ελήφθησαν ήταν έκτακτη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα έρχεται να τα αναθεωρήσει. Ο νέος τρόπος λοιπόν συντονισμού και παρακολούθησης των προϋπολογισμών έχουν δώσει θετικά αποτελέσματα στον περιορισμό των ελλειμμάτων. Υπάρχουν όμως μερικοί μηχανισμοί όπως οι μηχανισμοί επιβολής κυρώσεων που δεν έχουν ακόμα εφαρμοστεί αλλά φαίνεται ότι συνεισφέρουν για μια υγιή και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση. Θα πρέπει να έχουμε ένα σύστημα που να λειτουργεί όμως και να μπορεί να συνεισφέρει ε, στην αποφυγή των σφαλμάτων του παρελθόντος. Ένα σύστημα που να επιτρέπει στα κράτη-μέλη να κάνουν τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις και την πολιτική τους για να συνεισφέρει επίσης στην ανταγωνιστικότητα, την απασχόληση και την ανάπτυξη. Δίνονται κίνητρα στις συστάσεις αναχώρα και αυτές θα πρέπει να ενισχυθούν ακόμα περισσότερο για να υπάρξει η απαραίτητη ευελιξία, ας πούμε, όταν είναι έκτακτες οι περιστάσεις και αν πρέπει κάτι να αλλάξει ε, δεν νομίζω ότι είναι σκόπιμο να αλλάξει ολόκληρο διότι θα διακυβευθεί η αξιοπιστία τους. Οι μικρές χώρες ε, θα πρέπει να σεβονται τα ίδια κριτήρια με τις μεγαλύτερες. Ε, θα ήθελα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όμως να εγγυηθεί ε, ότι όλα τα κράτη-μέλη συμμορφώνονται προς τους κανόνες. Ευχαριστώ πολύ κυρία Παύνοβα και τώρα η κυρία Γκίλ για 1,5 λεπτό. Σα uh, Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα επαναλάβω αυτά που είπαν οι συνάδελφοι ότι απαιτείται να βελτιωθεί και να αναθεωρηθεί η οικονομική διακυβέρνηση της Ευρώπης. Η ανακοίνωση της Επιτροπής είναι ένα πρώτο βήμα, αλλά είναι ένα μικρό βήμα. Πρέπει να τερματίσουμε τις πολιτικές λιτότητας. Απαιτείται να υπάρξει σημαντική αλλαγή και εμείς σαν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε την νομοθετική αρμοδιότητα θα φτάσουμε τα 35 εκατομμύρια ανέργους, πληθωρισμό, υψηλά ελλείμματα, υπερβολικά χρέη. Όλα αυτά δυστυχώς χειροτερεύουν και δεν βελτιώνονται. Φυσικά το έλλειμμα πρέπει να μείνει κάτω από το 3% αλλά παρόλα αυτά υπάρχουν και άλλα τα οποία θα πρέπει να γίνουν και όχι μόνο αυτό να επιδιώκουμε. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και ορισμένους κοινωνικούς δείκτες τι κάνουν τα κρατη για να αντιμετωπίσουν την φοροαπαλλαγή, τις, ε, ε, τι δυνατότητες εκπαιδευτικές μπορεί να έχουν διάφορες χώρες που αντιμετωπίζουν προβλήματα. Ε, όχι μόνο στοιχεία για το έλλειμμα και το χρέος. Νομίζω ότι είναι διασυνδεδεμένες οι οικονομίες μας και γι' αυτό απαιτείται μια καλύτερη διαχείριση της ευρωπαϊκής οικονομίας με ευέλικτο τρόπο. Η μεταρρύθμιση του εξαπλού και του διπλού πακέτου θα είναι μια καλή ευκαιρία έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποδείξει ότι παίρνει σοβαρά υπόψη τα συμφέροντα του Ευρωπαίου πολίτη. Γι' αυτό λοιπόν απευθύνω έκκληση στον Αντιπρόεδρο Ντομπρόφσκι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μην λειτουργεί σαν ένα απλό λογιστή. Ευχαριστώ κύριε Αγγέλ. Για δύο λεπτά η κυρία Τόμσκ. You have not the floor. Δεν έχετε πια το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Συμφωνώ με τη διαπίστωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και όλων εκείνων οι οποίοι λέγουν ότι τα προηγούμενα έτη η οικονομική διακυβέρνηση είχε περιέλθει σε αδιέξοδο. Και τα δύο αυτά μέτρα και οι δύο δέσμες μέτρων προσφέρουν μία διέξοδο από αυτό το αδιέξοδο στο οποίο είχαμε βρεθεί. Τώρα, αν θα είναι αυτό επιτυχές δεν μπορεί κανένας να το προβλέψει ακόμα. Πρέπει να πούμε ότι ε, ε, χρειάζεται επιγόντως ένας βαθύτερος έλεγχος των δημοσιονομικών των κρατών μελών. Οι κυβερνήσεις φέρονται παράλογα καμιά φορά. Και προτιμούν να ε, χαϊδεύουν τα αυτιά των ψηφοφόρων τους. Εκτός ε, λοιπόν από την οικονομική ισορροπία και τη διακυβέρνηση είναι σωστό που έχει διατηρηθεί ο έλεγχος και συμπεριλαμβάνει και κοινωνικά στοιχεία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι έχει κάνει 42 ελέγχους σε βάθους και έχει διαπιστώσει 5 ε, περιπτώσεις με παρατυπίες χωρίς όμως να λάβει μέτρα και κυρώσεις να επιβάλλει. Άρα γεννάται το νέο ερώτημα. Αρκεί μια απλή υπόσχεση μιας κυβέρνησης, εμπιστεύεται μήπως υπερβολικά της κυβερνήσης Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μήπως δεν ελέγχει το περιεχόμενο των ε, ε, όσων έχει υποσχεθεί μια κυβέρνηση και σε ό,τι αφορά την εφαρμογή. Ε, σε ό,τι αφορά δε τη χώρα μου, τη Σλοβενία, μπορώ να σας πω ότι διαπιστώνω από τον πίνακα στο παράρτημα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακολούθησε και πίστευσε μάλιστα τις ε, υποσχέσεις της Ρωμανικής κυβέρνησης. Κανονικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να δίνει μεγαλύτερη προσοχή ε, στην εφαρμογή όλων αυτών των μέτρων και στην ουσία και όχι μόνο ότι τάζουν οι κυβερνήσεις να κοιτάει. Και επίσης ο Πρόεδρος διακόπτει την ομιλήτρια για 1,5 λεπτό το λόγο έχει ο κύριος Λούντβικσον. Det är viktigt att vi är mycket noggranna i vår analys. Πρέπει να, προσέξουμε πολύ την ανάλυση που κάνω. στο πλαίσιο της εξάπτυχης και δίπτυχης δέσμης κανονισμών. Ε, να δούμε τι έχει γίνει μέχρι τώρα, αλλά και με την αξιολόγηση των ρυθμίσεων που υιοθετήσαμε για την αντιμετώπιση της κρίσης. Οι κανόνες χρειάζεται να τροποποιηθούν δεδομένες της κατάστασης. Πώς χρησιμοποιούνται οι κανόνες αυτοί. Νομίζω ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Πρέπει οι ρυθμίσεις να είναι ευέλικτες, ευφύης. Το πρόβλημα όμως είναι ότι δεν γίνεται και ευέλικτη η εφαρμογή αυτών των κανόνων. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν και κατά πόσον υπάρχει και ένα είδος ιδεολογικής ε, κοντοθωρίας που συνοδεύει την εφαρμογή αυτών των ε, κανόνων. Σίγουρα πρέπει να υπάρχουν κανόνες και μέτρα, αλλά θα πρέπει αυτοί να εφαρμόζονται. Έτσι θα βελτιωθεί η κατάσταση και θα έχουμε και επενδύσεις στις χώρες που τις χρειάζονται περισσότερο. Το πρόβλημα λοιπόν δεν είναι οι ρυθμίσεις αλλά η εφαρμογή τους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Λούτριξον. Και τώρα ακολουθεί η διαδικασία Κατζιάη, τις αυθόρμητες τοποθετήσεις. Δυστυχώς έχω λάβει διπλάσιες αιτήσει ε, από το χρόνο που έχουμε. Οπότε θα περιορίσω τον κατάλογο. Ο συνάδελφος Μπόγκοβιτς λοιπόν πρώτος. Ε, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η Οικονομική και Δημοσιονομική Ένωση είναι πάρα πολύ σημαντική και για τις μεγάλες και για τις μικρές χώρες το ευρώ είναι από τις σημαντικότερες κινητήριες δυνάμεις ε, για μικρά ε, κράτη που προσανατολίζονται στις εξαγωγές όπως είναι η Σλοβενία. Ε, συμφωνώ με τους αυστηρούς κανόνες και συμφωνώ να ισχύουν και για μικρές και για μεγάλες χώρες. Επειδή έχουν αλλάξει οι συνθήκες, μετά από την οικονομική κρίση. Χαίρομαι για τη νέα δέσμη που προτείνει πλέον ο κύριος Γιούνκερ, από τη μια επιτρέπει αποτελεσματική ε, πολιτική με νέα μέτρα για δημιουργία θέσεων εργασίας, ε, με δημοσιονομική σταθερότητα αλλά και κοινωνικό κράτος. Γι' αυτό είμαι πεπισμένος ότι οι χώρες θα πρέπει να ελέγχονται πάρα πολύ προσεκτικά και πάρα πολύ αυστηρά για να εφαρμόζονται οι μεταρρυθμίσεις και μάλιστα ε, ιστοδυνικές. Και μακροπρόθεσμα οι μεταρρυθμίσεις είναι απαραίτητες για τις ίδιες τις χώρες, όχι μόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ο κύριος Πυρίνσκι. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Υπάρχουν ενδιαφέροντα στοιχεία στην παρουσίαση την οποία κάνατε. Στόχος του νέου μηχανισμού είναι να ενισχύσει υποτίθεται την οικονομική διακυβέρνηση έτσι ώστε να διασφαλιστεί ε, ασφάλεια, συνοχή και οικονομική ανάπτυξη. Νομίζω ότι η μεταβατική αυτή έκθεση στην ουσία δείχνει ότι θα πρέπει εμείς να φέρουμε πιο κοντά ε, τους ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης στα διάφορα κράτη-μέλη. Αυτό είναι όμως κάτι το οποίο ακόμα το επιδιώκουμε, δεν το έχουμε πετύχει. Και δεν υπάρχουν σε καμία περίπτωση στατιστικά στοιχεία τα οποία να αποδεικνύουν ότι θα πετύχουμε τους συγκεκριμένους στόχους. Τι ε, απαντήσεις μπορείτε να μας δώσετε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πυρίνσκι. Ο κύριος Μαριάς παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, από τη συζήτηση που έχει διεξαχθεί αποδείχθηκε ότι το τεράστιο δημοκρατικό έλλειμμα που ισχύει κατά τη διαδικασία της περίφημης οικονομικής διακυβέρνησης είναι δεδομένο. η επιτροπή χωρίς δημοκρατική νομιμοποίηση θεωρεί ότι μπορεί να καθορίζει την οικονομική και κοινωνική πολιτική των κρατών μελών θεωρεί ότι μπορεί να ελέγχει τους εθνικούς προϋπολογισμούς και να επιβάλλει στα εθνικά κοινοβούλια τι να πράξουν. μάλιστα ο κύριος juncker έχει εντελώς αποθρασινθεί και ενεργώντας ως εκπρόσωπος των δανειστών και της τρόικας παρεμβαίνει παράνομα στις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις στην ελλάδα στηρίζοντας τη μνημονιακή συγκυβέρνηση και τα μνημονιακά κόμματα εν ώψη των επικείμενων εθνικών εκλογών. το ίδιο κάνει και στην αθήνα τα τελευταία 24 ώρα ο κύριος μοσκοβισή. Κύριε της κομισιόν παρανομείτε και παραβιάζετε τη συνθήκη που σας επιβάλλει πολιτική ουδετερότητα. συμμαζευτείτε! να ξέρετε ότι δεν μπορείτε να τρομοκρατήσετε τον ελληνικό λαό που στι επικείμενε εκλογέ θα σα βγάλει κόκκινη κάρτα και θα σα στείλει το μήνυμα που σα αρμόζει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Μαριά. Και τώρα ο κύριος Γλέζος παρακαλώ. Υπάρχει μια αρχαία ελληνική παροιμία η οποία λέγει «Όδιν εν όρος και έτε κεν μην». Κυλοπονούσε το βουνό και γέννησε ένα ποντικό. Η εξάπτυχη και δίπτυχη δέσμη οικονομικών μέτρων δεν κατάφερε ούτε να γεννήσει ένα ποντικό. Δεν σταμάτησε τη λαιλασία του λαού υπέρ των τραπεζών. Δεν σταμάτησε την ανεργία στην Ελλάδα. Δεν σταμάτησε το κλείσιμο των μικρών επιχειρήσεων. Δεν σταμάτησε τη φτώχεια και την πείνα. Δεν σταμάτησε τις αυτοκτονίες. Αυξήθηκε το χρέος ακόμα πιο πολύ. Γιατί διότι στηρίζεται στη θεοποίηση του χρήματος, στην αντίληψη ότι το χρήμα παράγει τα πάντα. Μέγα λάθος. Το χρήμα αντιπροσωπεύει και ανταλλάσσει αξίες, δεν παράγει αγαθά. Αξίες και αγαθά παράγει μόνον ο εργαζόμενος με την εργασία του. Υπάρχει μια έρευνα ειδικών επιστημόνων που λέει ότι αν δεν υπήρχε η καταλήστευση της υπεραξίας των εργαζομένων αν δεν υπήρχαν τα προβλήματα τα εργατικά Ευχαριστώ κύριε συνάδελφε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Γιλέζο. Η κυρία Μάλετιτς. Ευχαριστώ πολύ Κύριε Πρόεδρε, να καλωσορίσω τον κύριο Ντομπρόφσκη και να τον συγχαρώ για την ε, αναφορά που μας έκανε. Θέλω να πω και εγώ ότι όπως και οι συνάδελφοί μου υποστήριξαν Πρόκειται για μια στρατηγική, συνεκτική, συντονισμένη προσέγγιση σε ό,τι αφορά την οικονομική διακυβέρνηση. Άρα είναι καλά αυτά τα μέτρα. Όμω πρέπει να αφήσουμε περιθώριο στα κράτη-μέλη ώστε να βρουν τι ε, βέλτιστε λύσει για τη δική του περίπτωση. Για τη μεσονομική σε διαθροτικέ μεταρρυθμίσει, επενδύσει. Δεν υπάρχει λύση αντιγραφή επικόλυση, copy-paste στην προκειμένη περίπτωση. Βέβαια μπορούν να ανταλλάσσουν εμπειρίες και να μαθαίνουν από τις βέλτιστες πρακτικές άλλων τα κράτη-μέλη. Όμως για ε, πέραν μάλλον των μεταρρυθμίσεων πρέπει και σε επίπεδο ένωσης ε, να προωθηθούν μεταρρυθμίσεις όπως για την κοινή αγορά, την ενία ε, την πολιτική συνοχή μεταξύ άλλων για να δημιουργηθεί μια ανταγωνιστική καινοτόμως Ευρώπη με μια οικονομία που θα ανακάμπτει και θα γίνεται όλο και πιο ισχυρή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ Μάρετιτς. Η κυρία Ρωσιάρ τελευταία για το ΚΑΤΣΙΑΙ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Όταν ε, ε, υπάρχουν δυσκολίες εύκολα βρίσκει κανείς τον αποδιοπομπαίο τράγο και μπορούμε να δείξουμε και μια διανοητική οκνηρία. Μιλάμε για την οικονομική διακυβέρνηση. Σίγουρα ε, δεν πρέπει να καταφύγουμε σε εύκολες λύσεις. Ε, με τον αποπληθωριστική αυτή περιδίνηση ε, όλοι θα παρασυρθούμε ανεξαρτήτως εθνικότητας. Πρέπει να γίνουν δημοκρατικές, δημοκρατικοί διάλογοι. Η ο στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε βέβαια μια πραγματικό νομική διακυβέρνηση που θα μας ε, θυμίσει αυτό που δεν πρέπει να πάψει να είναι η Ένωση, δηλαδή ε, ένα συνεργατικό σχέδιο, ε, δηλαδή κράτη που συνεργάζονται στην υπηρεσία του πολίτη. Και γι' αυτό βέβαια χρειάζεται αναθεώρηση των φυστάμενων μέτρων και εργαλείων και αυτό περιμένουμε από την Κομισιόν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κυρία συνάδελφε, κυρία Ροζιέ. Ολοκληρώνεται η διαδικασία ΚΑΤΣΙΑΙ και μετά για να κλείσει τη συζήτηση τώρα δίνω το λόγο στον Επίτροπο. Κύριε Ντομπρόφσκης, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Να σας ευχαριστήσω όλους για τη συζήτηση την οποία είχαμε σήμερα. <clears throat> Όπως είπα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί τις δυνατότητες ενίσχυσης και βελτίωσης της οικονομικής διακυβέρνησης και κομβικός μας εταίρος είναι πάντα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σημειώσαμε όλες τις προτάσεις σας και σημειώσαμε επίσης και τους, ε, τις περιοχές τις οποίες πολλά μένει να γίνουν ακόμα. Ευχαριστούμε την κυρία Μπερές και του Σκιώδης για τις παρατηρήσεις τους στα πλαίσια και της δικής τους έκθεσης ιδίας πρωτοβουλίας. Έγιναν και άλλες παρατηρήσεις, οι οποίες κάποιες από αυτές είναι εκτός της εμβέλειας, της αναθεώρησης του ΣΥΚΣΠΑΚ και του ΤΟΥΠΑΚ, της εξάπτυχης και της δίπτυχης δέσμης σχετικά με την καλύτερη χρήση σαν παράδειγμα της ευελιξίας Ξέρετε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προετοιμάζει μια λεπτομερέστερη ε, καταγραφή των δυνατοτήτων σωστότερης χρήσης της ευελιξίας στα πλαίσια του εξαπλού και του ε, διπλού πακέτου. Θα παρουσιάσουμε το έγγραφο αυτό ε, αρκετά νωρίς το 2015. Θα λάβουμε υπόψη μας τα θέματα τα οποία τέθηκαν και από σας όπως η λήψη υπόψη των οικονομικών κύκλων, ε, το θέμα της επένδυσης, το θέμα των διαρθαπτικών αλλαγών. <clears throat> Πάντως για μια ακόμη φορά θα πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι εμείς προετοιμάσαμε το κείμενο αυτό στο υπάρχον πλαίσιο ε, του πακέτου ειδικότερα το θέμα της αντιμετώπισης των επενδύσεων και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο για Στρατογικές Επενδύσεις είναι κάτι το οποίο έχει ήδη παρουσιάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, τέτοιου είδους επενδύσεις θα αντιμετωπιστούν ευνοϊκά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όλες τις άλλες δαπάνες οι οποίες έχουν σαν σχέση ή έχουν σαν στόχο μάλλον <clears throat> τη μείωση του χρέους και την τόνωση της ανάπτυξης και δεν θα δώσουν χώρο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προχωρήσει σε λήψη μέτρων. Θα υπάρξει δηλαδή μια ευνοϊκή μεταχείριση των χωρών οι οποίες κάνουν βήματα στον τομέα αυτό. Δεν έχει φυσικά τελειώσει η προσπάθεια ενίσχυσης γενικότερα του οικονομικού ευρωπαϊκού πλαισίου και νομίζω ότι τους επόμενους μήνες θα έχουμε πολλά να ανταλλάξουμε γύρω από τα θέματα αυτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ντομπρόφσκη, κύριε Πίτροπε. Ολοκληρώνεται λοιπόν εδώ η συζήτηση και διακόπτω τη συνεδρίαση μέχρι τις ψηφοφορίες.